Uh, good afternoon, everybody. Um, καλωσορίζω όλους. Έχουμε καθυστερήσει κατά 10 λεπτά. Από ό,τι φαίνεται έχουμε διαφορετικές ζώνες ωραρίων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη λοιπόν είναι η υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις ως προς αυτό. Μετά έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 26ης-27ης Ιανουαρίου του 2010 και της 22 και 23 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να σας πω είναι να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους Πολωνούς μέλη της Επιτροπής μας που είτε είναι παρόντες είτε μας ακούν σχετικά με το φοβερό δυστύχημα του Σαββάτου που οδήγησε στο θάνατο και τον Πολωνό Πρόεδρο αλλά και ε, πάρα πολλά στελέχη της πολιτικής ζωής της χώρας. Εις ένδειξη σεβασμού λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να σηκωθούμε και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Thank you. Uh, right, I, now continue. Θα συνεχίσω λοιπόν με τις ανακοινώσεις μου πριν περάσουμε στο workshop που θα ακολουθήσει. Να σας θυμίσω καταρχάς ότι την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεχίσουμε με την ακρόασή μας για τα μαθήματα στα οποία μπορεί να καταλήξει κανείς για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Η συνεδρίαση θα γίνει στο ημικύκλιο από τις 3 μέχρι τις 6.30. Έχω προσκαλέσει <clears throat> τους ομιλητές σε αυτήν την ακρόαση να κάνουν σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις για να υπάρχει χρόνος ερωτήσεων. Ας προσπαθήσουμε εμείς να συντονίσουμε τη φύση των ερωτήσεών μας θα σας στείλουμε ένα σημείωμα από τη γραμματεία. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να συμβουλέψω τα μέλη και τους συντονιστές <clears throat> ότι θέλουμε περιορισμό του χρόνου ομιλίας σε ένα λεπτό και θα πρέπει οι ερωτήσεις μάλλον να είναι ενός λεπτού και να είναι σε ένα συγκεκριμένο θέμα και όχι πολλαπλές αλλά αυτά θα τα αποφασίσουμε αφού συζητήσω λίγο σύντομα με τους συντονιστές στο τέλος της συνεδρίασης αυτής. Τέλος, σχετικά με τον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Χριστοδούλου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ευαίσθητη θέση στην οποία βρίσκεται ως υπεύθυνος της υπηρεσίας, της ελληνικής υπηρεσίας χρέους της ελληνικής δημοκρατίας και αύριο ξέρετε θα, ζητη, θα εκδοθεί ένα νέο ομόλογο από την Ελλάδα οπότε προφανώς είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η επόμενη συνάντηση 14 Απριλίου μετά τη Δευτέρα του Στρασβούργου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 Πέμπτη στο Στρασβούργο από τις 9.30 μέχρι τις 11.30. Συγγνώμη που έχουμε δύο συναντήσεις στο Στρασβούργο, αλλά αλλιώ δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες. Μετά 26 Απριλίου από τις 3 μέχρι τις 6.30. Τρίτη 27 από τις 9 το πρωί μέχρι το 6.30 το απόγευμα με το μεσημεριανό διάλεμα Όλα αυτά θα σας τα στείλουμε γραπτά. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε απευθείας στο workshop. Δεν γίνεται συνήθως ε, τέτοιου είδους συναντήσεις στις κανονικές συναντήσεις της Επιτροπής μας. Συνήθως γίνονται θα έλεγα ακροάσεις και τα λοιπά, μπορέσαμε να βρούμε αυτό τον χώρο και το χρόνο και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε για τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των οχημάτων, μηχανοκίνητων οχημάτων. τις επιπτώσεις των προτάσεων στους καταναλωτές, τους εμπόρους λιανικής και τους κατασκευαστές και την επίπτωση των νέων ρυθμίσεων για τις τιμές, τελικές τιμές τους καταναλωτές και την κατάσταση του ανταγωνισμού πριν από τις 31 ε, Μαΐου του 2013. Βλέπετε εδώ ότι έχω και τον πρόεδρο τον Μάλκομ Χάρμπορ της Επιτροπής ΣΥΝΚΟ. Υπάρχουν θέματα που άπτονται άμεσα των συμφερόντων των καταναλωτών, οπότε η παρουσία του εδώ και η εμπειρογνωμοσύνη του η προσωπική θα είναι πολύτιμη. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, περνώ στους ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο Πολ Τσίτσαρ. υπεύθυνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και του δίδω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μέλη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Κομισιόν στη σημερινή συνεδρίαση. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας όπως ήμασταν και στο παρελθόν για να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Τα μηχανοκίνητα είναι πολύ σημαντικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας και χρειάζονται αυτή τη στιγμή αναδιάρθρωση όχι μόνο λόγω της κρίσης αλλά και λόγω της υπερβολικής παραγωγής και της ανάγκης να παραχθούν πρασινότερα οχήματα. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο εδώ. Στον τομέα υπάρχουν από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου αλλά και χιλιάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο κατασκευαστών αλλά κυρίως ε, διαφόρων γκαράζ επισκευής. Επομένως για μας το σημαντικότερο θέμα είναι να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό αναλάβαμε μία μελέτη από το 2006 και κάναμε μία αποτίμηση το 2008. Πέρσι το καλοκαίρι κάναμε μία ανακοίνωση για τα συμπεράσματα της μελέτης και της αξιολόγησης και μετά και μόνο θεώρησε η Κομισιόν ότι μπορούσε να υποβάλει τις προτάσεις αυτές μετά από βέβαια δημόσια διαβούλευση. Οργανώθηκαν και δύο στρογγυλές τράπεζες με ενδιαφερομένους και δύο συνεδριάσεις Συμβουλευτικής Επιτροπής με εκπροσώπους των χωρών μελών το ΕΚΟΣΟΚ, γενικά υποστήριξη της προτάσεις μας και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και καταναλωτριών επίσης η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στον τομέα αυτών, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελε η Κομισιόν να εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει για διαφοροποιημένα, διαφοροποιημένα μάλλον μέτρα ανατύπου οχήματο. Εμείς θα θέλαμε να πούμε ότι ως προς τη μορφή της πρότασης προβλέψαμε καταρχήν μια γενική εξαίρεση βάσει της οποίας μόνο το 2013 θα αρχίσει να ισχύει το νέο καθεστώς για να μπορέσουν να τελειώσουν οι ισχύουσες επενδύσεις. Και άλλες αλλαγές έγιναν ως προς την αρχική πρόταση όπως η υποχρέωση πιστοποίησης των νέων κινητήρων και οι κανόνες διαφάνειας. Όπως συμβαίνει συχνά σε διαβουλεύσεις, η Κομισιόν δεν κατάφερε, δεν μπόρεσε να δεχτεί όλα τα σχόλια που ακούστηκαν, ιδιαίτερα δύο για τους ε, πολιτές. Για το λεγόμενο multi-branding θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό δεν έχει δημιουργήσει ούτε ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε ταραχή, ούτε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όσο για την προστασία των διαφόρων συμβολέων και συμφωνιών, δεν νομίζουμε και αυτό ότι είναι θέμα που μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει και το θέμα της σύνδεσης των θεμάτων αυτών με τις τελευταίες προτάσεις, σχετικές προτάσεις του Συμβουλίου, τις οποίες η Κομισιόν δέχεται. Και όπως οι περισσότεροι από τους ενδιαφερομένους και εμεί θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία να αποσαφινιστεί το νομικό πλαίσιο τώρα για να υπάρχει στο μέλλον νομική βεβαιότηση. Έχουμε μοιράσει και ορισμένα τυπωμένα, ορισμένες τυπωμένες διαφάνειες να μπορείτε να τις κοιτάξετε για να καταλάβετε καλύτερα την διαδικασία αυτή. Δεν έχουμε προβολέα βέβαια. Α, ε, έχουμε. έχουμε. Τέλεια. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε ότι βλέπετε λέγω ότι η γενική εξαίρεση που προβλέψαμε, block exemption, είναι κάτι για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα για να προστατεύσει τα ενδιαφερόμενα μέρη από έρευνες αντιτράστα αλλά χωρίς να καθορίσει τι ακριβώς είναι καλή και κακή συμπεριφορά και αντιανταγωνιστική. Δεν καθορίζει δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρότυπο, απλώς περιγράφει. Στη δεύτερη διαφάνεια βλέπετε ότι ήδη από το 2006 θελήσαμε να αναλάβουμε μια μελέτη η οποία έδειξε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα των νέων αυτοκινήτων, αλλά υπάρχουν προβλήματα στην αγορά και η πώληση των υπολείπων των παλαιών αυτοκινήτων δηλαδή, και για πολλούς λόγους θεωρήσαμε ότι η πρωτογενής αγορά έχει σωστές συνθήκες ανταγωνισμού. Υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτήν και πέφτουν οι τιμές και όλα αυτά δείχνουν ότι έχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα ο τομέας. Κατά τα υπόλοιπα δηλαδή τον μη πρωτογενή τομέα υπάρχουν θέματα κατάχρησης των εγγυήσεων ή έλλειψης πρόσβασης στην απαραίτητη τεχνική πληροφόρηση κλπ. Και ανταλλακτικά. Προτείναμε αλλαγές στην ε, εξαίρεση που καθορίσαμε γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι το απαραίτητο αλλά όχι επαρκές. Τώρα, πώς θελήσαμε να γίνει, να διευκολυνθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών ή να επιτραπεί στους ε, επιδιορθωτές η πώληση εναλλακτικών ανταλλακτικών και να εφαρμόζονται με τα νενομισμένα δίκτυα οι εγγυήσεις. Η ευθυγράμμιση με τους ισχύοντες κανόνες είναι η κύρια προσέγγισή μας. Δεν θεωρούμε ότι στην πρωτογενή αγορά ή τμήμα του τομέα χρειάζεται καμία πρόσθετη νομοθεσία. Ούτε αλλάζει τίποτα ως προς την υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για την πώληση από παράλληλα δίκτυα. Και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και τα μέρη της ε, βιομηχανίας συμφώνησαν. Όσο για τις ισχύουσες, ε, για τους ισχύοντες του multi-branding, θεωρούμε ότι οι κατασκευαστές που είχαν εκφράσει το φόβο ότι θα αλλάξει η εικόνα που έχουν στην αγορά οι διάφορες γνωστές μάρκες έχουν καθησυχαστεί. Το multi-branding που είναι θέμα που πολλοί το συζήτησαν και αμφισβήτησαν, θα συνεχίσει να επιτρέπεται στις αγορές γιατί είναι θέμα αγοραστικής, ε, αγοραστικού ρεαλισμού ή ρεαλισμού της αγοράς. Διότι η παραγωγή οχημάτων εξαρτώνται από τους διανομής σε, σε πολλά μεγάλα αστικά κέντρα και πρέπει να μπορούν ορισμένοι πολιτές που να, έχουν το δικαίωμα να πολλούν διάφορες μάρκες, ιδιαίτερα σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Και το αντίθετο τώρα το single branding δηλαδή. Ας μην σας διαβάσω ακριβώς τι λέει η αφάνεια, μπορείτε να το διαβάσετε. Το 2 κοιτάξτε ιδίω, γιατί και το 4 που προέκυψαν από τις συζητήσεις μας με τους ε, πολιτές, τους οποίους ακούσαμε προσεκτικά γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι φραγμός στην πολιτική του ανταγωνισμού μια ευθυγραμμισμένη πολιτική επιβολή των κανόνων και υποστηρίζουμε και μια δεοντολογία την οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι πολιτέ διότι μόνο έτσι θα υπάρξουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ κατασκευαστών και πολιτών. Τώρα για τα συμβόλαια. Σας τα είπα αυτά που λέει η διαφάνεια και προηγουμένως. Θα τόνισα ιδιαίτερα ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι τα προβλήματα των πολιτών, θεωρητικά ή πραγματικά, πρέπει να λυθούν είτε εθνικά, από εθνική νομοθεσία, είτε ενωσιακά μέσω τροποποίησης της σχετικής οδηγίας. Αν έχετε απορίες θα μπορώ να σας τις λύσω, αλλά γενικά δεν θεωρούμε ότι η πολιτική του ανταγωνισμού μειώνει σε τίποτε την ε, ικανότητα των πολιτών για διαπραγμάτευση. Τέλος, θεωρούμε ότι η πρόταση θα ενδυναμώσει τον τομέα που αφορά πάρα πολλές θέσεις εργασίας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και νομίζω, όπως και οι συνάδελφοί μου, ότι η νέα προσέγγιση καταλήγει σε καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του τομέα. Είναι βασικό οι κατασκευαστές να έχουν το δικαίωμα πιο αποτελεσματικά να καθορίζουν τα δίκτυα πώλησης και ο ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτών και μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών να παραμείνει ζωντανός. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μάρκ Γκρέβεν, Διευθυντής της Υπηρεσίας Νομικών Υποθέσεων για τους αυτοκινητοβιομηχάνους. Νομίζω και αυτός έχει διαφάνειες ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής, ε, να σας παρουσιάσω την άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Αυτοδιογενείας για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανευθέωση της γενικής αυτής εξαίρεσης. Ε, με δύο λόγια, η άποψή μας είναι ότι η Κομισιόν υπέβαλε μια καλή πρόταση από το έργο που επιτέλεσαν βλέπουμε ότι η αγορά της αυτοκινητίας οπωσδήποτε είναι εξίσου ανταγωνιστική, αν όχι περισσότερο ανταγωνιστική, όπως άλλες αγορές άλλων προϊόντων. Και γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κανένας λόγος να διατηρήσουμε πιο περιοριστικό νομικό πλαίσιο για το δικό μα τομέα σε σχέση με άλλου τομείς το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε αυτό τον κανονισμό γενικών εξαιρέσεων και στο δικό μας τομέα. Παραδεχόμαστε βέβαια ότι ίσως υπάρχει νόημα να διατηρηθούν ορισμένοι ιδιάζοντες κανόνες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό αφορά την αδιαθυσμότητα των αναλλακτικών και την δυνατότητα επισκευής που είναι πιο σημαντική στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας από τις άλλους τομείς. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το δεχτούμε και θα θέλαμε οι νέοι κανόνε να εφαρμοστούν το φλεγόρατο των δυνατών. Με γενικέ γραμμέ όσον αφορά την ε, αγορά που ακολουθεί την αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική. 50% είναι ανεξάρτητη και εμεί έχουμε το 50% και γι' αυτό δεν έχουν κανένα πρόβλημα για τη διατήρηση ορισμένων συγκεκριμένων κανόνων για τα ανταλλικά, για τι εγγυήσει και επίση για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών για την ε, συντήρηση και τι επισκευέ. Και σήμερα οι αυτοβιογανοί θα εξακολουθούν να διαθέσουν, διαθέτουν συγγνώμη, αυτές τις πληροφορίες για όλα τα οχήματα που βρίσκονται στην αγορά. Το κάνουμε, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και επίσης για τα πιο σύγχρονα οχήματα, αυτά που είναι σύμφωνα δηλαδή με τα πιο πρόσφατα πρότυπα εκπομπών, το Ευρω 5 δηλαδή για τα επιβατικά αυτοκίνητα και το ε, Ευρω 6 για τα επαγγελματικά. Αυτό είναι ένα όρο για την έγκριση τύπου. Αν δεν διαθέτουμε δηλαδή αυτέ τις πληροφορίες δεν μπορούμε να πάρουμε την έγκριση τύπου. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει εδώ κάποιο πρόβλημα και δεν περιμένουμε να υπάρχουν σημαντικέ επιπτώσει για ιονδήποτε στον τομέα αυτό τη αγορά κατόπιν τη πώληση του οχημάτου. Όσον αφορά τώρα τι ε, πωλήσει των οχημάτων, σα είπα ότι βρισκόμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση όπω και στι άλλε αγορέ προϊόντων πολύ ανταγωνιστική αγορά, δεν υπάρχουν ειδικά προβλήματα. Είχαμε κάποια ειδικά προβλήματα την τελευταία φορά που η Κομισιόν αναθεώρησε του κανόνε γενικών εξαιρέσεων, γιατί υπήρχαν τότε κάποιε διαφορετικέ τιμών και ήταν δύσκολο οι αγοραστέ να αγοράζουν τα προϊόντα σε μια άλλη αγορά και ορισμένοι μάλιστα υπέστησαν πρόστιμα ε, από την Κομισιόν γιατί πουλούσαν τα αυτοκίνητά τους σε διαφορετικές τιμές, αλλά από το 2005 και μετά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε, είναι ότι αν εφαρμόζουμε αυτή τη γενική εξαίρεση, δεν θα σημαίνει αυτό ότι θα αλλάσουν τα πάντα. Μάλλον όταν κινηθούμε από το σημερινό κανονισμό στο γενικό κανονισμό, δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις καθόλου. Λίγα σημεία νομίζω Ίσως αξίζει να αναφέρουμε εδώ σχετικά, γιατί κατά τα άλλα τα πράγματα θα παραμείνουν λίγο πολύ όσοι έχουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι αν κάποιος σας πει ότι αυτή είναι επανάσταση, δεν πρέπει να το πιστέψετε. Δεν είναι σωστό. Πού θα έχουμε διαφορές από τους κανόνες, τους καινούργιους, όπως είπε και ο είναι στον τομέα του λεγόμενου multi-branding. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν έμπορο που πουλάει διαφορετικές, ε, διαφορετικών εταιριών αυτοκίνητα. Αυτό υπάρχει εκεί που έχει ένα νόημα οικονομικά, παραδείγματο χάρη σε ε, αγροτικές ε, περιφέρειες, όπου δεν υπάρχει κανένα νόημα ο κάθε κατασκευαστής να έχει για τη δική του μάρκα ένα κατάστημα, αυτό θα αυξήσει μόνο περιτά το κόστος. Λοιπόν, η multi-branding θα υπάρχει πάντα παντού όπου είναι οι προϋποθέσεις κατάλληλες. Το άλλο σημείο που να αναφέρουμε είναι οι συμβατικές ε, ρήτρες, όπως τις λέει η Κομισιόν, ή ορισμένοι το αποκαλούν σαν ε, τα θέματα που προστατεύουν τους ε, εμπόρους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό Είναι ένα πραγματικό θέμα, υπάρχουν θέμα, αλλά όχι ένα θέμα που αφορά τον ανταγωνισμό. Ε, μετά έχουμε το δικαίωμα του εμπόρου να πουλήσει το κατάστημά του σε κάποιον άλλον. Η πολιτική λέει ότι αν κάποιο θέλει να σταματήσει τη δραστηριότητε θα πρέπει να προειδοποιήσει δύο χρόνια προηγουμένως και να καταγγείλει τη σύμβαση που υπήρχε. Και εκεί που υπάρχουν προβλήματα θα μπορεί να υπάρχει διατησία και να μην χρειάζεται άμεση προσφυγή στο δικαστήριο. Γιατί το δικαστήριο και πιο ακριβό είναι και πιο χρονοβόρο. Αυτά κατά γνώμη δεν είναι θέματα ανταγωνισμού, δεν έχουν επιπτώσεις στον καταναλωτή ή στην προσφορά του προϊόντος ή στην τιμή των αυτοκινήτων. Αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με τον ανταγωνισμό. Είναι θέμα συμβατικών σχέσεων. και ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτό αναγνωρίζεται γιατί αν δει κανένα και άλλου τομεί γενική εξαίρεση, όπω τη γενική γενική εξαίρεση, βλέπετε ότι δεν αναφέρεται τίποτα για προστασία του πιο αδυνάμου μέρου στου κανόνε αυτού, παρόλο που αφορά παραδείγματο χάρη τι ε, ελληνικές λιανικέ προπολίσει τροφίμων. Και όλοι συμφωνούμε νομίζω ότι τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο ισχυρά από τις εταιρείες από τις οποίες αγοράζουν τα προϊόντα τους. Παρ' αυτά κανένας δεν θεώρησε ότι θα έπρεπε να ε, προτείνει κανόνες που θα προσπαθεύουν εκείνους από τους οποίους τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν. Γιατί λοιπόν να το έχουμε εδώ. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιους κανόνες. Και επίσης άλλος κανόνας που δεν χρειαζόμαστε είναι εκείνος που δίνει το δικαίωμα στους εμπόρους να πουλήσουν την επιχείρησή τους το σε επιχείρηση είναι, αλλά είναι και η μάρκα του κατασκευαστή που εκπροσωπείται. Και γι' αυτό, εάν πρέπει να απολυθεί ε, ένα κατάστημα, θα πρέπει και ο, ο κατασκευαστής να έχει λέγην. Να υπάρχει δηλαδή για μια συναλλαγή μεταξύ του κατασκευαστή και του εμπόρου. Και αυτή ήταν η κατάσταση πριν από το 2002, πριν έχουμε δηλαδή τον τρέχοντα κανονισμό και θα πρέπει νομίζω να επανέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Και γιατί γιατί είδαμε με τον ισχύοντα κανονισμό κάποιες καταστάσεις που νομίζουμε ότι δεν είναι προς όφελος του κοινού. Είδαμε μεγάλες ομάδες εμπόρων, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αγόρασαν άλλους, συνήθως με δανεισμένα χρήματα φυσικά, και μετά με την οικονομική κρίση, αυτές οι ομάδες βρέθηκαν σε δυσκολίες, όπως και άλλες ε, επιχειρήσεις γενικά, και το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισαν να κλείνουν διάφορα καταστήματα, διάφορες αντιπροσωπείες και ο κατασκευαστής έμεινε με το πρόβλημα στα χέρια του και ορισμένες ε, μεγάλες περιφέρειες αγροτικές ιδίως έμειναν χωρίς εκπροσώπηση της συγκεκριμένη μάρκας. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Από την άλλη μεριά όταν συζητάμε στην ελάχιστη περίοδο καταγγελίας, η δυνατότητα διατησίας, αν υπάρχει κάποια διαμάχη για τη σύμβαση, Πιστεύουμε ότι αυτό είναι θέμα καλών επιχειρησιακών πρακτικών. Θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά εκτός του κανονισμού. Είναι κάτι που θα πρέπει να συμφωνθεί μεταξύ των ε, συμβαλλαγμένων μερών. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστέ, οι Ιάπωνε κατασκευαστέ υιοθέτησαν κανόνα συμπεριφορά στα πλαίσια του οποίου έχουν αναλάβει την ε, υποχρέωση να διατηρηθούν τα δύο αυτά σημεία στι συμφωνίε για τι αντιπροσωπείες και θα μπορούν επίσης να προασπιστούν τα σημεία αυτά στο δικαστήριο. Τα έχουν δηλαδή τα δικαιώματα που έχουν και σήμερα οι ε, αντιπρόσωποι. Τέλος, όσον αφορά τη χρονική στιγμή θέση ισχύω των νέων κανόνων. Ξέρουμε ότι η πρόταση είναι να αναβληθεί η εφαρμογή των κανόνων πώληση μέχρι το 2013. Εμεί πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να εφαρμοστούν αμέσω όπως και στους κανόνες για την αγορά κατόπιν πόλης του οχήματος, γιατί και στις δύο περιπτώσεις θα ήταν πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστούν και στον τομέα των ε, πωλήσεων και στον τομέα των υπηρεσιών ήδη κανόνες την ίδια χρονική στιγμή. Αν δεν γίνει θα είναι ατυχές. Θεωρούμε ότι η αναβολή αυτή δεν είναι πολύ χρήσιμη γιατί έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση οι πωλήσει αυτοκινήτων μέχρι τα τέλη του έτου έχουν πέσει κατά 20% σχέση με το 2007, οι πωλήσει ε, φορτηγών κατά 35% και κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να προσαρμόσουμε την ε, κατασκευαστική βιομηχανία τις αντιπροσωπείες και δεν έχουμε χρόνο απεριόριστο μπροστά μα. Αυτό που θα να τονίσω σήμερα είναι να συστήσω σε όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν την απόφαση για το μέλλον του κανονισμού για τη γενική εξαίρεση το γλυγορότερο δυνατόν και να μην αναβάλουν τίποτα. Πολλά έχουν αναλυθεί, όλα έχουν αναλυθεί. Έχουν γίνει πάρα πολλέ μελέτε για τι επιπτώσει και αν δεν ληφθεί η απόφαση τώρα, η βιομηχανία αυτή θα είναι σε μεγάλη βεβαιότητα μέχρι το 2013, χωρί να ξέρει τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Και αυτό κατά τη γνώμη είναι το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Και οι περισσότερε ανταγωνιστικέ αρχέ συμφωνούν με την Κομισιόν. Η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή συμφωνεί επίση με την πρόταση και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε μια ομιλία σε δύο τμήματα από τους Ρόμπινσον και Σάιξ. Δεν ξέρω ακριβώς τι κατανομή χρόνου έχετε κάνει μεταξύ σας, δεν ξέρω καν ποιος θα ξεκινήσει, έχετε το λόγο πάντως, η κυρία Ρόμπινσον. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να υπογραμμίσουμε τις απόψεις των εμπόρων. Εκπροσωπούμε 380.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη με 2.800.000 υπαλλήλους μικρομεσαίες επιχειρήσεις η διεύρυνση μέχρι το 2013, η παράταση ήταν κάτι το θετικό. Από την άλλη είμαστε απογοητευμένοι από τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Αν δούμε τι έχει πετύχει μέχρι τώρα η παρούσα εξαίρεση, έχει επιτρέψει τη λειτουργία την διασυνοριακή της αγοράς, έχει επιτρέψει το multi-branding, έχει επιτρέψει τη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης των εμπόρων και αυτό είναι κάτι που βοήθησε τους εμπόρους ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ύφεση. Αυτό ωφελεί τον καταναλωτή και σε επίπεδο επιλογής και σε επίπεδο τιμής. Δίδει επίσης τους εμπόρους την δυνατότητα να επενδύσουν, την εμπιστοσύνη να επενδύσουν και σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μία μέση επένδυση 2,5 με 3 εκατομμύρια αναμονάδα. Ταυτόχρονα δίδει στους καταναλωτές τη δυνατότητα σύγκλησης των τιμών, τους δίνει μεγαλύτερη επιλογή, διαθεσιμότητα των οχημάτων, η εμπιστοσύνη των εμπόρων λοιπόν έχει τονωθεί, δεν θα λειτουργούσαμε σωστά χωρίς τα συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε την δυνατότητα να πολλούμε, να αλλάζουμε ιδιοκτησίες, έχουμε τη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία. και ελέγχεται μερικές φορές το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων εμπορικών, εμπορίας αυτοκινήτων εννοούμε πάντα βέβαια, ε, για να δούμε αν δεν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κινήσεων που μπορεί να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία για τις συγκλήσεις των τιμών. Προφανώς δεν είναι το μοναδικό ε, ενδιαφέρον παράδειγμα, αλλά παρουσιάζει συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Το νέο σύστημα δυστυχώς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χαλαρό. Ο κανονισμός ε, ο ισχύων είναι 88 σελίδες και είναι αρκετά χρήσιμος για τους εμπλεκομένους. Αλλά υπάρχει μία αύξηση των σελίδων σε 146 σελίδες με πάρα πολλά εκτελεστικά μέτρα και ερμηνευτικές διατάξεις και δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο θεωρείται βελτίωση της νομοθεσίας. Στην ουσία βάζει ξανά σε ηγέτιδα θέση τους κατασκευαστές και βάζει στην ίδια κατηγορία την αγορά αυτοκινήτων με την αγορά καλλιντικών προϊόντων κτλ. Είναι υπερβολική η νομοθεσία. Η ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στους κατασκευαστές και τους εμπόρους ήταν κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και ευαίσθητο. Η Επιτροπή θέλει ένα πάρα πολύ ε, εξαδυνικευμένο θα λέγαμε οικονομικό πρότυπο δεν αναγνωρίζει την ανισότητα μεταχείρισης ανάμεσα στους κατασκευαστές και τους εμπόρους και αυτό φύγει τους καταναλωτές. Ο κανονισμός που ισχύει σήμερα ε, έκανε βήματα προόδου για την αποκατάσταση της ισορροπίας. Όλα αυτά τα μέτρα δυστυχώς χάνονται. Αυτή η πολύ θεωρητική αντιμετώπιση του θέματος ε, θα θίξει τον καταναλωτή, θα υπάρξει έλλειψη επιλογής, έλλειψη ανταγωνισμού τέλος θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο ασθενής πήρε το φάρμακο, φαίνεται ότι βελτιούται η κατάστασή του, οπότε ας τον σταματήσουμε, να μην παίρνει πλέον το φάρμακο αυτό, μιας και πάει καλύτερα. Συνεχίζει η κυρία Σάιξ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Θα ασχοληθώ με τα θέματα που έχουν σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίο προωθούν οι οργανώσεις των παραγωγών όπως επίσης και το θέμα του εάν η επανεξιολόγηση των συνθήκων ανταγωνισμού στην βασική αγορά πρέπει να γίνει πριν από το 2013 ή έστω και μετά το 2013. Θεωρούμε σαν οργάνωση των εμπόρων <coughs> ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία της εξουσίας αν θέλετε ανάμεσα στους καταναλωτές και τους εμπόρους. Μέχρι τώρα τα πράγματα είχαν βελτιωθεί μέχρι τώρα έτσι ώστε να έχουν οι έμποροι αυτοκινήτων ε, την ικανότητα να αντέξουν στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές πιέσεις ε, στις οποίες τους εκθέτει η ελευθερία μέσα στην οποία λειτουργούν. Multi-branding, διασυνοριακές πωλήσει, δυνατότητες εισαγωγής ευθυνότερων ανταλλακτικών, ανεξαρτησία προμηθευτών, όλα αυτά λειτουργούν διασυνοριακά. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να εφαρμοστούν ε, στον καινούριο κανονισμό έτσι όπως προτείνεται. Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό λοιπόν να εγκαταλείπονται όλα αυτά τα μέτρα στο όνομα δήθεν της ναι, καλύτερης νομοθετικής ρύθμισης δίδεται πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους κατασκευαστές ότι δεν θα ασκήσουν την εξουσία τους εις βάρος ε, των εμπόρων και αντίθετα από αυτά που μας είπε ο κύριος Γκρέβεν στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στον τομέα χονδρικής και στα σούπερ μάρκετ ε, οι αρχές ελέγχου του ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κάνουν κάτι μετά από 10 χρόνια αρπακτική συμπεριφορά των μεγάλων εταιριών και κατανοούν ότι οι εθελοντικοί κώδικες δεν λειτουργούν όταν υπάρχει μια τόσο έντονη ανισότητα στην ισορροπία ανάμεσα στους εμπόρους και τους ε, κατασκευαστές έτσι ώστε ε, να προστατευτούν και οι καταναλωτές. Έχουμε λοιπόν παράλληλα τέτοια συστήματα να συγκρίνουμε ανάμεσα στον δικό μας τομέα και τον τομέα των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Οι κατασκευαστές είναι σε θέση να ασκούν τεράστια πίεση στις εμπορίες αυτοκινήτων, όχι μόνο διαπραγματευόμενοι τους όρους, αλλά και μέσω άλλων συστημάτων όπως τα μπόνους, όπως των απειλών για λήξη και ε, απαγόρευση ανανέωσης, αδειοδότησης πώλησης και ε, ε, πρόορης διακοπής των συμβάσεων αν ένας έμπορος πιέζεται και άλλος ένας έμπορος πιέζεται να μην αγοράσει έναν μικρότερο έμπορο κάτι το οποίο του φαίνεται σαν σωστή επιχειρηματική κίνηση, τότε δημιουργούνται προβλήματα στρέβλωσης των ανταγωνισμού και χάνεται η επενδυτική δυνατότητα. Οι νέες ρυθμίσεις λοιπόν που προτείνονται για το 2013 δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη στην εμπορία αυτοκινήτων και αυτά είναι άσχημα νέα για όλους όσους επιθυμούν καλύτερες υπηρεσίες στον τομέα προστασίας του καταναλωτή και όχι αποκλειστικής προστασίας του κατασκευαστή. Ένας κώδικας συμπεριφοράς μπορεί να είναι χρήσιμος, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα μεταφοράς και να ελέγχει τους τρόπους και τις αιτίες διακοπής συμβάσεων από πλευράς των κατασκευαστών. Διαφωνούμε λοιπόν με τις απόψεις που ακούστηκαν νωρίτερα ότι ε, τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι συμβατές με τον ισχύοντα νομικό, με τον ισχύοντα νομικό, ε, το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τώρα για την αξιολόγηση των συνθήκων ανταγωνισμού. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ήταν σημαντική, έγιναν τεράστιες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκομένους, αλλά τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κυκλοφόρησαν πριν από το Μάιο του 2008, πριν ολοκληρωθεί δηλαδή η προσπάθεια αξιολόγησης. Βασίστηκαν στις πληροφορίες που είχαν συλλέξει από το 2002 μέχρι το 2006 αυτό ήταν μια κίνηση θα έλεγα ανώριμη και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεψε να ληφθούν υπόψη τα ωφέλη των νέων ελευθεριών τις οποίες είχαν στη διάθεσή τους οι έμποροι αυτοκινήτων. Πάρα πολλά θα έλεγα στοιχεία ισχύοντα σήμερα στην αγορά αυτοκινήτων και στην εμπορία αυτοκινήτων τέθηκαν σε ισχύ δύο χρόνια μετά από την εξέταση αυτών των στοιχείων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα μάλιστα βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες χωρίς προηγούμενο ίσως στη διεθνή οικονομία και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα επιπλέον. Υπάρχουν 4,3 νέοι αγοραστές αυτοκινήτων που προχωρούν στη συγκεκριμένη αγορά και είναι περίεργο να βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις από τη μία τους οδήγησαν στο να κάνουν την αγορά τους και από την άλλη τεχνητά να αποσυνδέουν την αγορά αυτή από την ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων. Συνεπώς λοιπόν ε, οι αγορές αυτές, οι οποίες μάλιστα γίνονται κατά 80% από ε, πρόσωπα άνω των 60 ετών και ε, μάλιστα και από πρόσωπα τα οποία πολλές φορές δεν είχαν αγοράσει μέχρι τώρα αυτοκίνητα. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ εύθραυστη, η κατηγορία αυτή των αγοραστών είναι πάρα πολύ ευάλωτη, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα δίκτυα αυτοκινήτων που αγοράζουν τα οχήματά τους και θέλουν να τους αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα. Συνεπώς οι πιέσεις τις οποίες ασκούν οι κατασκευαστές μετά την αγορά είναι κάτι το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο ε, τις δυνατότητες και τα ωφέλη των νέων αυτών καταναλωτών. Εν πάση περιπτώσει δεν θα περάσω στις λεπτομέρειες της επόμενης διαφάνειας, αλλά θα πρέπει η αγορά αυτή να γίνει αντικείμενο επαναξιολόγησης πριν το 2013. Φοβάμαι ότι αν τυχόν δεν υπάρχει πλέον τροχοπέδη σε αυτήν την πορεία, οι συνέπειες θα είναι άσχημες για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο οποίος θα μας παρουσιάσει ε, την άποψη των καταναλωτών. Κρίντ. Σας ευχαριστώ κύριε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να μιλήσουμε και εμάς. Θέλω να σας πω ποιος είμαι. 79 εθνικές ε, ε, ομάδες αν προσωπούμε στην Ευρώπη και ασχολούμαστε με τα προβλήματα των καταναλωτών ασχολούμαστε μόνοι του τους κατανοητές. Σε κάθε βήμα ε, δίνουμε συμβουλές με τα περιοδικά μας, βοηθάμε τους κατανοητές όταν έχουν ε, κάποια βλάβη στην άκρη του δρόμου, απαντούμε σε ερωτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά τις επισκευές και τις συντηρήσεις των οχημάτων. Είμαστε λοιπόν πραγματικά μια οργάνωση για τους κατανοητές, ειδικευμένη στους ε, Κινητικού καταναλωτέ. Βλέπετε λοιπόν ότι αναγνωριζόμαστε στον ρόλο μας αυτό μέσα της ε, διαδικασίας και του κανονισμού 1400 του 2002. Εργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια της ε, Στρογγυλή τράπεζα τη ομάδα υψηλού επίπεδου με την Επίτροπο κυρία Κρού και τώρα είμαστε η μόνη φωνή που εκπροσωπεί τους καταναλωτές στη διαδικασία αυτή. Επιπλέον έχουμε δράσει έντονα, έντονα με τους ε, ενδιαφερόμενους για τον τομέα της ε, αυτοβιομηχανίας και βρισκόμαστε εδώ για να εξετάσουμε τις πτυχές ε, του καταναλωτή στη συζήτηση. Βλέπετε εδώ για τους καταναλωτές καταρχήν το αυτοκίνητο είναι η δεύτερη πιο σημαντική δαπάνη ενός νοικοκυριού μετά από ένα σπίτι. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι ε, με τη διάρκεια των ετών η συντήρηση και οι επισκευές κοστίζουν εξίσου όσο η αρχική αγορά του οχήματο. Αυτό είναι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αγαθό και γι' αυτό χρειάζονται ειδικοί κανόνες για την αγορά αυτή. Μέχρι στιγμής υπάρχει ε, έλλειψη ενιαίας, ενιαίου διακονισμού της ε, πρωτογενούς αγοράς και της αγοράς κατόπιν της πόλης του οχήματος. Βέβαια, ε, υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν δυσνόητες διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός, μικρότερη επιλογή και θα αυξηθεί και η τιμή. Θα ήθελα να τονίσω και μια άλλη πτυχή. Γενικά, υπάρχουν περισσότερες επιλογές κινητικότητας, όχι μόνο όσον αφορά το αυτοκίνητο, αλλά και το θέμα της υπηρεσίας για ένα και χρονικό διάστημα της ελεύθερης ε, επισκευής. Είναι δύσκολο λοιπόν οι καταναλωτές να καταλάβουν όλες τις επιλογές που υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο multi-branding που και η Κομισιόν και όλοι οι άλλοι εμβαλόμενοι και ενδιαφερόμενοι τόμισαν ότι θα αλλάξει σημαντικά τις προτινόμενες διατάξεις. η συγκέντρωση στην πρωτογενή αγορά θα σημαίνει για τους ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο για να οργάσουν τα οχήματα. Θα είναι πιο δύσκολη σύγκριση, γιατί παρόλο που είναι δυνατή να γίνει σύγκριση των τιμών σε διάφορα επίπεδα, παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο είναι κάτι που θέλει κανένα να δοκιμάσει. Θέλει να δοκιμάσει διάφορε μάρκε του ίδιου προϊόντος. Και αυτό θα πρέπει η αγορά να είναι σχετικά κοντά στην κατοικία του καταναλωτή. Το multi-branding επέτρεψε σε νέες μάρκες όπως το Kia να επικρατήσουν σε αγορές που κατά τα άλλα δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αν δεν είχε αυτή η δυνατότητα. Και θέλω επανέλθω σε ένα από τα επιχειρήματα που άκουσα από τους προαλήσαντες. Η κατάσταση πραγματικά βελτιώθηκε από το 2002. Εξοδόμαστε των καταναλωτών θα ανησυχούσα να αλλάξει το σύστημα που είδαμε ήταν πολύ θετικό για τους καταναλωτές. Στην ε, λεγόμενη αγορά κατόπιν της του οχήματος βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φορές ε, προβλήματα για την ε, εγγύηση που δίνεται κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί περισσότερο το θέμα του multi-branding και να ξέρουμε ότι η αλληλή των κανόνων θα οδηγήσει ενδεχομένω σε μια μείωση του ανταγωνισμού και να είναι ει του καταναλωτή. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο θέμα σημαντικό για μας, το θέμα των ε, εγγύησεων. Όπως βλέπετε υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσει. Υπάρχει η νόμιμη εγγύηση και η ε, εκεί. Η Κομισιόν ε, θεωρούσε ότι υπήρχαν προβλήματα νομισμού γιατί ορισμένοι από του κατασκευαστέ τείνουν η διευρυμένη εγγύηση να ε, είναι συνδεμένη με αποκλειστική επισκευή του οχήματος υπό του, του αρχικού πολιτή. ότι αυτό θα μείωνε τον οργανισμό και τις τελικές επιλογές του καταναλωτή. Εδώ βλέπετε ότι η τρέχουσα πρόταση Κομισιόν είναι να εξτάσει το θέμα της εγγύησης κατευθύνες γραμμές και να δει ότι αυτό δεν καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα των εγγύσεων, αν παραδείγματος ένας ε, κατασκευής ε, δίνει δωρεάν συμπληρωματική εγγύηση για επισκευές ή για συντήρηση. Εμείς ενισχύουμε γιατί αυτό δεν αναφέρεται στην ε, εγγύηση, γιατί είπαμε ότι αυτό δεν θα αφορά όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά θα είναι χαρακτηριστικό για όλους τους κατασκευαστές γιατί τονίζει τι χρειάζεται και τι γίνεται και πιστεύω ότι αυτή η εγγύηση θα πρέπει να συμπεριλάβατε στο mini BR. θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί και το θέμα αυτό στη μελλοντική νομοθεσία και να δώσει δυνατότητα ο καταναλωτής να μπορέσει να κάνει την καλύτερη επιλογή για τον ίδιο και να μην είναι δεσμευμένο για κάποια συγκεκριμένη μάρκα ή κάποιο δίκτυο. Επίσης λέγεται ότι θα θέλουν οι καταναλωτές λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά για να αγοράσουν το αυτοκίνητό τους. Μπορεί αυτό να είναι αλήθεια, αλλά δεν θα θέλουν να πάνε 100 χιλιόμετρα για να αλλάξουν ένα λάστιχο. Αυτό είναι κάτι που μας ενδυχεί. Και τέλος, πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο και χρήσιμο για να υπάρχει μια ανταγωνιστική αγορά και δεν μπορούν να γίνουν επισκευέ χωρίς να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Και εδώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα από τα επιχειρήματα των συναδέλφων της ΕΣΕΑ που είπαν ότι οι ίδιες πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται και στους ε, αντιπροσώπους και στις ε, δευτερεύουσες ε, αγορές και σε εκείνους που επισκευάζουν ενδεχομένω αυτοκίνητα. Αυτό όμως δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε αναγκαμένοι να πάμε να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν κάποια βλάβη και βλέπουν ότι οι προφορίες δίνονται σε διαφορετικά διαφορετικές μορφές και οι πληροφορίες που χρειάζεται το κάθε μέσα πρέπει να δίνεται ακόμα και αν ε, περνάει πέρα τα όρια εκείνα που έχουν εκείνοι που είναι διακριμένοι από τις αντιπροσωπείες. Οι πρόοδο λοιπόν στις τεχνικές ε, πληροφορίες, εμείς θέλουμε τα ίδια, όπως και η Κομισιόν. Θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα αυτό και θα πρέπει να είναι κύριο τμήμα που θα συμπεριλαμβάνεται στο mini BR. Αυτό αναφέρεται εδώ και στι κατευθυντέ γραμμέ που θα είναι δεσμευτικέ. Το κατάλαβα με αυτό που το είπε η Κομισιόν, αλλά πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα συμπληρωθούν με μια αναφορά αυτών στο MiniBR. Και θεωρούμε επίση ότι πλήρης ορισμός των τεχνικών πληροφοριών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο φάκελο των Ευρω 5 θα πρέπει να προσθεθεί στο MiniBR. Με δύο λόγια λοιπόν, αυτό που η θέλει σαν εκπρόσωπε από τον καταναλωτών είναι να εξασφαλιστεί ο καταναλωτής στην αγορά μετά την πώληση και τα χρόνια μέχρι το 2013 να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί το multi-branding για να δούμε κατά πόσον υπάρχει καλύτερος τρόπος διακανονισμού μετά το 2013 και να υπάρχει πλήρης ορισμός το τι σημαίνει πρόσβαση στις ε, τεχνικές πληροφορίες και αυστηρή διατάξη όσον αφορά τι εγγυήσει και την πρόσβαση στι τεχνικέ πληροφορίε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική προσφορά για του καταναλωτέ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αρχίσει ο γύρος των ερωταπαντήσεων αλλά και η συζήτηση. Ο Μάρκολ είναι ήδη έτοιμος και γι' αυτό θα μιλήσει πρώτος. Αν θέλει άλλο το λόγο να το ζητήσει. Παρακαλώ. Ορίστε. Σας κατευχαριστώ Σάρα. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και σας και την Επιτροπή σας για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης και για την ευκαιρία που μας δίνεται να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για αυτά τα θέματα. Όπως είπατε και προηγουμένως, έχει υπάρξει, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον επανειλημμένο στην Επιτροπή μας για τέτοια πληροφόρηση και γι' αυτό θα ήθελα να θέσω μόνο μερικά και συγκεκριμένα ερωτήματα, στοχευμένα. Το ενδιαφέρον μας για προβλήματα των καταναλωτών είναι προφανές φάνηκε και από όσα ακούσαμε σήμερα. Γι' αυτό θα ήθελα να δηλώσω πριν θέσω ερωτήματα ότι ορισμένες αρκετές οργανώσεις καταναλωτών έχουν επίσης υποβάλει αιτήματα στην Κομισιόν για τα θέματα ακριβώ που συζητήσαμε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω τώρα είναι λίγο γενικό, λίγο όμως. Ε, και θα ήθελα να το σχολιάσει η Κομισιόν αλλά ίσως και οι άλλοι ομιλητές. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, συμμετέσχον και εγώ σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μακροχρόνια συζήτηση, για την παρατήρηση των εξελίξεων στον τομέα που έδειξαν από τα δεδομένα που συνελέχθησαν ότι η μελέτη υπήρξε επιτυχής. Πρώτα απ' όλα, οι πολιτές έκαναν, είπαν κάτι σημαντικό, δηλαδή ότι η ανάλυση της στρατηγικής της Κομισιόν διατυπώθηκε πριν να σημειωθούν οι τελευταίες και αξιοσημείωτες αλλαγές στην αγορά. Ερωτώ λοιπόν, σε τι στοχεύει η αλλαγή αυτή. Οι καταναλωτές δεν ζήτησαν αλλαγή, ούτε κατασκευαστές. Και από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει και καμία σημαντική οικονομική λειτουργία που να δικαιολογεί αλλαγή. Με βάση ποιο δημόσιο ενδιαφέρον λοιπόν ή συμφέρον διατυπώνεται η πρόταση αυτή. Αυτό το ερωτώ προς την Κομισιόν βέβαια. Δεν κατάλαβα καθόλου σε τι θα ωφελήσει τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες η πρόταση αυτή. Αυτό ήταν το πρώτο μου ερώτημα, γιατί πολιτικά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει όντως πραγματικά δημόσιο ενδιαφέρον και συμφέρον εδώ πριν συζητήσουμε. Στην παρουσίαση της Κομισιόν άκουσα κάτι που θα ήθελα να μου εξηγηθεί για τις ισχύουσες λέει πρακτικές του multibranding που θεωρεί η Κομισιόν ότι βλάπτουν και τους καταναλωτές και καταναλώτριες και τους πολιτές και πολίτριες. Θα ήθελα να γνωρίζω γιατί οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα. Καλό θα ήταν νομίζω οι καταναλωτές και οι πολιτές να έρθουν να μας πούν τι φρονούν ακριβώς για αυτή την πρακτική της πώληση διαφόρων μαρκών, multibranding. Για να μάθουμε κι εμείς Ποιο είναι ακριβώς αυτό το περίφημο δημόσιο συμφέρον. Και τέλος, η τεχνική πληροφόρηση. Καταρχήν νομίζω ότι οι εγγυήσει που ζητάει η Κομισιόν για τις πωλήσει παλαιότερων αυτοκινήτων, το λεγόμενο aftermarket δηλαδή, είναι κάτι ενδιαφέρον μεν, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω για την τεχνική αυτή πληροφόρηση που φαίνεται, μου φαίνεται ότι είναι κάτι ζωτικότατο. Όπως είπε σωστά η Κομισιόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει νομική υποχρέωση και ένα συγκεκριμένος ορισμός περί του τι είναι, τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτή η υποχρεωτική τεχνική πληροφόρηση και τα συζήτησε αυτά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να μου σχολιάσει λοιπόν η Κομισιόν εάν πράγματι πιστεύει ότι η έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών, γιατί νομίζω αυτό κάνανε και όχι κάποια σοβαρότερη νομοθεσία, αν οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν είναι τίποτα που θα διασφαλίσει ότι η τεχνική πληροφόρηση που απαιτείται για αυτοκίνητα που δεν καλύπτονται από την οδηγία του 2009 πρόκειται να εφαρμοστεί. Διότι από τις κατευθυντήριες γραμμές διαβάζω ότι το άρθρο 101 που αφορά τον ανταγωνισμό δεν, και το ξαναλέω, δεν εφαρμόζεται για την υποχρέωση χορήγησης τεχνικής πληροφόρησης. Ενώ ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν για την πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι και ακριβώς το γεγονός ότι η πληροφόρηση καμιά φορά χορηγείται με τέτοια μορφή που είναι άχρηστη τελείως. Ενώ για τα καινούργια αυτοκίνητα έχει καλυφθεί το θέμα. Από ό,τι λέτε όμως για τα παλαιότερα δεν θα υπάρχει αυτή η νέα μορφή πληροφόρησης. Εξηγήστε μου λοιπόν Πώς θα διασφαλίσετε ότι η τεχνική πληροφόρηση θα δίνεται στο ίδιο επίπεδο και για τα καινούργια και για τα υπάρχοντα αυτοκίνητα. Πώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σιλβί και μετά οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε άλλη. Αλλιώς θα ζητήσω τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση έχει σχέση με αυτά που είπε ο Μάλκο Μάρμπορ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αιτία των αλλαγών στις οποίες προχωρήσατε. Υποστηρίζετε ότι υπάρχουν λόγοι για την αλλαγή της νομοθετικής ρύθμισης, αλλά δεν τους βλέπουμε τους λόγους αυτούς. Δεν είστε πιστικοί. Αν κάτι πρέπει να αλλάξετε δεν θα έπρεπε να έχει σαν στόχο την ενθάρρυνση νέων τύπων παραγωγής αυτοκινήτων πιο πράσινων. Ο κύριος Μπαρόσο αυτό εκφράζει δημόσια. Πρέπει να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες εξηγήσεις και τότε μόνο θα σας ακολουθήσουμε, λέει η κυρία απευθυνόμενη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε τέτοιες ερωτήσεις όλοι ίσως μπορεί να κληθούν να δώσουν μία απάντηση. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν το πάνελ με τη σειρά με την οποία πήραν το λόγο. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δίνεται τη δυνατότητα να απαντήσω, λέει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τι τεχνικά στοιχεία και πληροφορίε για το λεγόμενο aftermarket μετά την πώληση. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν ήταν επαρκείς. Εμείς στοχεύουμε να ελέγχουμε την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων. Ξέρετε ότι το 2007 προχωρήσαμε σε διώξεις εις βάρος ε, τεσσάρων μεγάλων κατασκευαστών για τη μη κυκλοφορία των τεχνικών στοιχείων που απαιτείτο. Mm. Συνεπώς λοιπόν ότι πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός βασίζεται σε έλεγχο κατά περίπτωση και όχι σε υπερβολική νομοθετική δραστηριότητα. Τα λεγόμενα hardcore δηλαδή ε, είναι στην ουσία κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία, αλλά είναι πανάκια για τα προβλήματα. Δυστυχώς οι απλές νομοθετικές διατυπώσεις από μόνες τους δεν ικανοποιούν πλήρως τις επιθυμίες μας. Πρέπει να επιβάλλουμε και να ελέγχουμε την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών και γι' αυτό εμείς μέσω των ρυθμίσεων αυτών, ακόμα και αν φαίνονται πιο περίπλοκε, θα διευκολυνθεί ο έλεγχός μας. Και θα υπάρχει και πολύ καλύτερη ενημέρωση σε επίπεδο τεχνικό στα πλαίσια του λεγόμενου aftermarket. Είναι σαφές ότι θα πρέπει οι κατασκευαστές να ε, υπακούσουν, να σεβαστούν τις ρυθμίσεις αυτές Γιατί αλλαγές, η τελευταία ερώτηση. Ίσως να με συμπληρώσουν εδώ οι συνάδελφοι, αλλά θα έλεγα ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε πεπισμένοι ότι στα πλαίσια του aftermarket ο καλύτερος έλεγχος, ο πληρέστερος έλεγχος είναι προαπαιτούμενος. Υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα τα οποία μας ζητούν να τα αγοράσουμε με τις διαφημίσεις, αλλά το θέμα είναι όταν αγοράζουμε αυτοκίνητο μετά από δύο χρόνια να πηγαίνουμε να κάνουμε μία αλλαγή, μία επισκευή και αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτά πρέπει να τα ελέγξουμε και πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης και γι' αυτό προτείνουμε τις αλλαγές αυτές στο λεγόμενο aftermarket σχετικά με την πρωτογενή αγορά. Οι έρευνες που ξεκινήσαμε το 2006 αποκαλύπτουν ότι υπήρξαν επιπλέον κόστη τα οποία υφίσταντο οι έμποροι. Στην ουσία τα περνούσαν τα κόστη αυτά οι <clears throat> κατασκευαστές στους εμπόρους, στην εμπορία αυτοκινήτων και με τον τρόπο αυτό έλεγχαν τους εμπόρους για να αποτρέψουν το λεγόμενο multi-branding. Και αυτά τα κόστη φυσικά πέρναγαν στο τέλος τον ίδιο τον καταναλωτή. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι κατασκευαστές αυτή τη στιγμή θα είναι ηγέτες. Ξέρουμε τα προβλήματα υπερχωρητικότητας που έχουν στις διαδικασίες παραγωγής, ξέρουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, τη δυσκολία πώλησης αυτοκινήτων και έτσι οι κατασκευαστές θέλουν να έχουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά δίκτυα πώλησης και διανομής τα οποία να είναι οικονομικά όσο περισσότερο γίνεται για τους καταναλωτές και εκεί παρεμβαίνουμε. Πιστεύουμε ότι καθιστώντας το σύστημα στην πρωτογενή αγορά πιο ευέλικτο και οι έμποροι και οι κατασκευαστές από κοινού θα μπορέσουν <clears throat> να διανύμουν τα προϊόντα τους αποτελεσματικότερα. Ξέρετε ότι μερικές φορές το κόστος αυτό της διανομής είναι το 30% του κόστους του συνολικού ενός αυτοκινήτου για τον κατασκευαστή. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες και εκεί ακριβώς θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία προς όφελος της οικονομίας και των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Οι κατασκευαστές θα ήθελαν όχι. Σύντομα, δεν θα πω εγώ περισσότερο από άλλους το ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα το κάνει, αλλά η βιομηχανία πάντως θεωρεί, η άποψη της βιομηχανίας είναι ότι σήμερα σαν παραγωγικές επιχειρήσεις ελεγχόμεθα από έναν κανονισμό εξαίρεσης ο οποίος είναι λεπτομερής, δεσμευτικός ιδιαίτερα σε πάρα πολλούς τομείς από ότι οι γενικότερες ρυθμίσεις που αφορούν άλλους τομείς. <clears throat> Και δεν κατανοούμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί όπως σας είπαμε προηγουμένως, αν αναλύσει κανείς την αυτοκινητοαγορά, αγορά, δεν θα βρει να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα των πωλήσεων που δεν υπάρχουν σε άλλα προϊόντα. Το θέμα λοιπόν είναι η βιομηχανία να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο αντίστοιχο με τις άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν θέλουμε να διαφοροποιούμεθα από τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες. σχετικά με την αύξηση του κόστους. Αυτό ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αληθές. Εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ με μονομένους κατασκευαστές. Γνωρίζετε όμως ότι δεν έχουν ουσιαστικά πρόβλημα με το λεγόμενο multi-branding. <clears throat> Έχουν όμως πρόβλημα να πωλείται ε, το αυτοκίνητό τους παράλληλα με το αυτοκίνητο μιας άλλης εταιρείας μέσα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι αυτό που τους απασχολεί, δηλαδή στο κατάστημα δεν θέλουν να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος ε, για την πώληση των προϊόντων αυτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν να αποφύγουν οι ε, κατασκευαστές. Δεν είναι εναντίον του multi-branding πάντως γενικότερα. Κάποιοι από αυτούς έχουν θέσει και κάποιες, κάποιες απαιτήσεις για το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να βρίσκονται οι αντιπροσωπείες έτσι ώστε να μπορούν να πολλούν τα προϊόντα της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Μια τελική παρατήρηση για τη συντήρηση των αυτοκινήτων. Σε επίπεδο νομικό δεν υπάρχει καμιά διαφορά αν οι κανόνες αυτοί αποφασίζονται ε, σε επίπεδο κατευθυντηρίων γραμμών, κανονισμών, κανονισμών εξαιρέσεων. Το θέμα είναι να ελέγχονται οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται. Το είδαμε και στο παρελθόν. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει να υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο πληροφοριών για την επισκευή ας πούμε των αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει και θα χρησιμοποιήσει τα άρθρα που της δίνουν την δυνατότητα αυτή ε, στα πλαίσια όλων των νομικών βάσεων <clears throat> τις οποίες είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει. για την ενιαία φόρμα, για όλα τα αυτοκίνητα, για όλες τις βιομηχανίες. Είναι υποανάπτυξη στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπηρεσίας που ασχολείται με την εξομοίωση των ρυθμίσεων. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για την εφαρμογή του συστήματος αυτού στα παλαιότερα αυτοκίνητα. Ίσως να μην είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουμε εμείς στους επισκευαστές μας, ιδιαίτερα για αυτοκίνητα τα οποία παρήχθησαν εδώ και 10-15 χρόνια. Μερικές φορές δεν υπάρχει παρά μόνο ένα CD διαθέσιμο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα στο παρελθόν θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα στάνταρ τα οποία ισχύουν σήμερα. Υπάρχουν πληροφορίες, οι ανεξάρτητοι επισκευαστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά σήμερα και το ίδιο θα κάνουν και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους πολιτάς. Ευχαριστώ. Η Χίλαρη Σάιξ. Προς στιγμήν θα ήθελα να μιλήσω για έναν αριθμό μόνο που θεωρείται κάτι δεδομένο αλλά που ε, δεν είναι πια σωστό ότι 30% των οχημάτων της τιμής των οχημάτων οφείλεται στο κόστος της διανομής. Αυτά είναι πραγματικότητες του 99. Εγώ μαζί με άλλους πολιτές θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση των συνθήκων της αγοράς για να δούμε αν είναι αληθές αυτό, γιατί <laughs> φανταζόμαστε ότι δεν είναι πια. Για το multi-branding τώρα, μόνο δύο χρόνια ισχύει η άδεια αυτή για τους πολιτές να πουλούν πολλές μάρκες μαζί. και από ό,τι γνωρίζουμε από πρόσφατα στοιχεία του Νοεμβρίου και με παράδειγμα τη γερμανική αγορά, 68% των Γερμανών πολιτών πουλάνε διάφορες μάρκες ανακατεμένες. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι στα πλαίσια της κρίσης που γνωρίζουμε, είναι δε υπέρ του καταναλωτή. Πολλά από το πολλό μεγάλο μέρος του κόστους διαχείρισης, εγκαταστάσεων κλπ μοιράζεται το κόστος αυτό σε πολλά δίκτυα. Αν κανείς εκπροσωπεί δύο-τρεις μάρκες με το ίδιο σαλόνι ή με σαλόνια διαφορετικά με ένα αλλά κοντινά, αυτό σημαίνει ότι ως πολιτής έχετε καλύτερη προστασία από την κρίση. Γιατί έτσι το κόστος διαχείρισης για όλες αυτές τις μάρκες και τις πωλήσει των αυτοκινήτων τους συρρυκνώνεται. Τουλάχιστον μέχρι να διορθωθούν οι οικονομικές συνθήκες. Οι νέες όμως προτάσεις δεν θα καταλήξουν σε απλή επαναχώρηση κατά ένα βήμα, δηλαδή ότι θα ξανατεθούν διαχωριστικοί φραγμοί μεταξύ των μαρκών, αλλά δύο βήματα πίσω θα πάμε. Δηλαδή να διαχωρίζονται οι μάρκες και γεωγραφικά και νομικά ακόμα. Φανταστείτε πόση νομοθεσία θα χρειαστεί και τι γραφειοκρατικό βάρος θα χρειαστεί να φέρει μια επιχείρηση με αυτές τις προτάσεις, το οποίο βάρος θα περάσει ως κόστος βέβαια στους καταναλωτές. Τώρα, αν το multi-branding αύξησε το κόστος, πρέπει να γνωρίσουμε ότι σε κάποιο βαθμό ναι, γιατί οι κατασκευαστές θέλουν να διαφοροποιήσουν τη μάρκα τους λέγοντας ότι είναι καλύτερη από τις άλλες. Αλλά οι δυνάμεις της αγοράς είναι αυτές που καθορίζουν σε ποιο βαθμό μπορούν να επενδύσουν οι πολιτές για να αγοράσουν τα αυτοκίνητα που στη συνέχεια θα πουλήσουν δηλαδή. γιατί αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι οι καινούργιες μάρκες όπως η Hyundai αρχίζουν με πολύ χαμηλά πρότυπα και μετά τα αυξάνουν τις απαιτήσει τους για τον τρόπο πώλησης δηλαδή. Όταν όμως υπάρχει κρίση τότε συμφέρον θα είχαν όλες οι μάρκες να επιτρέψουν το multi που δεν μπορεί να το επιβάλλει στο κάτω-κάτω ο κατασκευαστής γιατί ο καταναλωτής και η καταναλώτρια θα καταλήξει τελικά να διαπιστώσει στη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή στην εξαφάνιση ορισμένων μαρκών από την περιοχή του. Τέλος, για το free riding. Αν βασιστούμε σε έναν αριθμό 2,5, μεταξύ 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ για το συνδυασμό των δραστηριοτήτων του πολιτή και του επιδιορθωτή. Τότε πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το κόστος επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Αυτό και αυτό μέρος του κόστους για τον πολιτή. Το multi-branding δεν είναι δικαιολογία για να καλυφθούμε πίσω από άλλα κόστη διότι ο πολιτής και όχι ο κατασκευαστής πρέπει να απορροφήσει το κόστος της διαχείρισης της επιχείρησής του. Το free riding μπορεί να αποφευχθεί μέσω μιας μικρής σύντομη περίοδου πώλησης μίας αποκλειστικά μάρκας, αλλά στη συνέχεια θα έπρεπε όλες οι υπόλοιπες μάρκες, όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστές δηλαδή, να δεχτούν ότι είναι συμφέρον των καταναλωτών και καταναλωτριών να έχουν μεγαλύτερη επιλογή μαρκών από το ίδιο σαλόνι. Γιατί αλλιώς ο κατασκευαστής τους επιβάλλει να αυξήσουν το κόστος της λειτουργίας της επιλογής τους αυτής. Ναι, η Κρίστα και μετά θα επανέλθουμε. Κυρία Κρίντ μάλλον. Για το multi-branding πάλι. Μπορεί να είναι πρόβλημα ότι ορισμένες μάρκες θα θεωρήσουν ότι δεν είναι πια τόσο ξεχωριστές αν πουλούνται μαζί με άλλες. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα ένας πολιτής να λειτουργεί διάφορα σαλόνια στο καθένα από τα οποία να πουλάει μία μάρκα. Υπάρχουν λύσεις. Με εκπλήσει που λέτε ότι αυξήθηκε το κόστος για τα καταναλωτή από το multi-branding, ενώ η Κομισιόν λέει ότι ελάχιστα συνέβη κάτι τέτοιο. Πρέπει να μάθουμε τους ακριβείς αριθμούς. Συμφωνώ ότι οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι δεσμευτικές και ότι από νομικής απόψεως είναι ισότιμες με το mini bear. θα μπορούσε η παραβίασή τους να οδηγήσει και σε προσφυγή στα δικαστήρια. Πράγμα το οποίο βέβαια θα αύξανε το κόστος λειτουργίας κάποιων μικρών αυτοκινηταγορών. Δεν θεω, λέω λοιπόν ότι δεν είναι η οι κατευθυντήριες γραμμές, αλλά ότι μπορεί από τη δεσμευτικότητά τους να επιβαρύνουμε το κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κλίμπ και Περές. Σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Αναφερθήκατε σε θέματα ανταγωνισμού, σε θέματα μείωσης του κόστους. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν προορισμοί σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ρύθμιση αυτή στην απασχόληση, στην παραγωγή και στη διανομή. Αν υπάρχει ανταγωνισμός υψηλός υπάρχει μείωση κόστους. Η μείωση κόστους θα πρέπει να προέλθει από κάπου. Θα ήθελα να μάθω ε, τι συνέπειες θα υπάρξουν στην απασχόληση. Θα ήθελα επίσης να μάθω τι συνέπειες μπορεί να έχουμε στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όταν μιλάμε σε, μεταξύ μας για τα θέματα αυτά, μία από τις δυνατότητες μείωσης του κόστους παραγωγής είναι η κυκλοφορία και η διάθεση προϊόντων που δεν είναι ε, τόσο καλής ποιότητας σαν τα αρχικά, τα πρωτότυπα θα έλεγα προϊόντα και αναφέρομαι κυρίως τα ανταλλακτικά. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασικά. και στην ουσία εντάσσεται στη λογική ε, του προηγούμενου συναδέλφου. Η Επιτροπή λειτουργεί συλλογικά όταν παρεμβαίνει σε ένα νομοθετικό τομέα, εντάσσει την νομοθεσία αυτή στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής που ακολουθεί. Και γι' αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει μια τριπλή διάσταση εδώ η οποία μας ενδιαφέρει. Ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής και διανομής υπάρχει το θέμα της υγείας γενικότερα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της, ε, της υψηλότερης παραγωγής από τη ζήτηση σε σχέση με την κρίση. Πώς οι ρυθμίσεις αυτές οι νομοθετικές θα επηρεάσουν την βιομηχανία αυτή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τελικά στη διάθεσή της έναν βιώσιμο τομέα και αποτελεσματικό τομέα. Η δεύτερη διάσταση είναι το θέμα της απασχόλησης πάλι. Καθένας από τους εμπειρογνώμονες αναφέρθηκε στη βασική ανησυχία την οποία έχει ο καταναλωτής. Στο σημερινό πλαίσιο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και εδώ έρχομαι και συμφωνώ με τον συνάδελφο Κλούντ, όταν μιλάμε για την αυτοκινητοβιομηχανία σκεφτόμαστε αμέσως την απασχόληση. Παράγονται τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από ένα πολύ ψηλό αριθμό εργαζομένων, ιδιαίτερα από περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μία μελέτη επιπτώσεων σχετικά με τις προτάσεις αυτές. Έχω μάθει ότι έχει κάνει, αλλά αυτό έχει γίνει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που είχε στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, ποιες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις. Το θέμα δεν είναι μόνο να αγοράζουν φτηνότερα αυτοκίνητα οι καταναλωτές, το θέμα είναι να δούμε πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν, πόσες θα χάσουμε και πώς θα τις διανύμουμε εδαφικά. Μία τρίτη ανησυχία μου παραπέμπει σε μία ερώτηση την οποία έχει ήδη γίνει αλλά δεν έχει τύχει απάντησης. Αν ελέγξει κανείς τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα και θα συμφωνήσετε μαζί μου, όλοι έχουμε ανησυχίες σχετικά με την αηφόρο ανάπτυξη. Ίσως αύριο να έχουμε ε, λιγότερα ιδιωτικά αυτοκίνητα, να υπάρχουν συλλογικότερε μορφές μεταφοράς και εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία να μολύνουν λιγότερο. Τι κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλοι δύο έχουν ζητήσει να θέσουν ερωτήσει. Ευχαριστώ ένα ερώτημα προς την Κομισιόν αλλά και προς τους ομιλητές. Οι αλλαγές που βλέπονται πώς θα επηρεάσουν μια χώρα με μικρό αριθμό διανομέων, υψηλή φορολόγηση των αυτοκινήτων, υψηλές τιμές καυσίμων και πολύ χαμηλό πληθυσμό, πολύ, πολλές αεροκατοικημένες περιοχές. Πώς θα επηρεάσουν οι αλλαγές αυτές λοιπόν τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες αλλά και τους πολιτές. Και εννοώ τη Φιλανδία, δηλαδή τη χώρα μου. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι αν οι πολιτές και οι πολίτριες δεν είναι σε θέση να πουλήσουν πολλές μάρκες μαζί, τότε οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες δεν έχουν ε, σύγκριση και επιλογή. Αν δυσκολευτεί το multi-branding θα χρειάζονται ορισμένοι να ταξιδέψουν μακριά για να δουν άλλες μάρκες από αυτές που θα πολλούνται τοπικά. Ο Ανδρέας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέρον το ερώτημα της κυρίας Σαγιά. δεν πρέπει νομίζω να τονίσουμε ιδιαίτερα μόνον τα οικοφιλικά αυτοκίνητα, τα περιβαλλοντοφιλικά αυτοκίνητα, αλλά να εξισορροπήσουμε τα συμφέροντα των κατασκευαστών από τη μία με δυνατότητα να ελέγχουν σε κάποιο βαθμό την αλυσίδα της διανομής, πράγμα που πειράζει και τις θέσεις απασχόλησης, με από την άλλη μεριά ε, τα συμφέροντα των πολιτών και διανομέων, διότι και αυτοί δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Τώρα το κατά πόσον μπορούν να επηρεάσουν τους κατασκευαστές συζητιέται. Λοιπόν, από την άποψη του καταναλωτή, όπως και ο Μάλκολμ Χάρμπουρ, δεν είμαι και εγώ πεπισμένος ότι ο κανονισμός του 2002 εξισορρόπησε τα πράγματα δεν εξισορρόπησε τα πράγματα ή ότι η τωρινή πρόταση θα είναι καλύτερη. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο και δεν με έπεισαν τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής. Γι' αυτό ερωτώ τον κύριο Γκρέβεν. Θεωρείτε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει η φυστάμενη ισορροπία με τις νέες προτάσεις ή μήπως ή μήπως λέγω από το 2011 και μετά τα μέτρα αυτά θα καταλήξουν να φανούν άδικα. Μάλιστα όλοι τώρα ξυπνάνε λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, έχω ακόμη τέσσερις ομιλητές. Ελπίζω να σημειώσατε. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Πρεσέδο. Μέχρι τώρα ο κανονισμός λειτουργούσε καλά. Χωρίς με τόσο σαφή διαχωρισμό μεταξύ πρωτογενούς τομέα και aftermarket. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καθαρά οικονομική πλευρά των πραγμάτων. Λοιπόν, οι σχέσεις δηλαδή μεταξύ κατασκευαστών και διανομέων. Αλλά και τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες πρέπει να δούμε. Τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά επί της τιμής για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Και η εξυπηρέτηση μετά την αγορά και η επιλογή τέτοιου είδους επιχειρήματα ενδιαφέρουν τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες η εφαρμογή των νέων αυτών νομικών προτύπων μπορεί να απαιτήσει τεχνολογικές αλλαγές. Νέα ανοιχτότερα δίκτυα ας πούμε. Πώς μπορεί το καινούργιο σύστημα να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές αλλαγές που ήδη διαπιστώνουμε. Η κυρία Ντάτη. Ευχαριστώ, εγώ θα είμαι συντομότατη. Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο το είχαμε συζητήσει το θέμα και πολλοί από εμά είχαν ζητήσει από την Κομισιόν να κάνει μια αξιολόγηση, μια μελέτη πολύ πιο συγκεκριμένη από τα πρώτα στοιχεία που μας είχε δώσει. Και βλέπω ότι δεν είναι πολύ συγκεκριμένη η μελέτη που έγινε ούτε για την απασχόληση ούτε για την κατανάλωση ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης. με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τα μέτρα στήριξης όπως το πριμ που δόθηκε για την απόσυρση και με το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς έχουμε εδώ τις μελέτες τις ίδιες, τις παλιές. Δεν λύθηκε το ερώτημα που είχαμε θέσει δηλαδή στην Κομισιόν, ιδιαίτερα ως προς την επίπτωση στην απασχόληση. Γιατί δεν, είναι το θέμα μόνο η κατανάλωση αλλά και η απασχόληση. Όπως είπε και ένας συνάδελφος δεν πρόκειται τα μέτρα αυτά να οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις. Μήπως κανείς άλλος ή καμία άλλη. Όχι. Τώρα θα απαντήσουν οι ομιλητές, αν και πολλές ερωτήσεις αφορούσαν την Κομισιόν. Σαφώς φαίνεται μάλλον πάντως ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για συζήτηση αυτού του θέματος πριν την προθεσμία που έχει τεθεί για την εφαρμογή των αλλαγών. Λοιπόν, ας με απαντήσει πρώτα η Κομισιόν λοιπόν. Έχουμε καμιά εικοσαριά λεπτά, πέντε λεπτά ο καθένας από τους απαντητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι που δεν είναι παρόντες σήμερα και που θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει και αυτή στη συζήτηση. Το θέμα είναι πολύπλοκο, το είχαμε δει και τον περασμένο Οκτώβριο. Είδατε ποιες είναι οι μελέτες μας. Έχουμε προχωρήσει και σε μελέτες επιπτώσεων επίσης. Υπάρχει μία τέτοια μελέτη πολύ σημαντική η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές και αξιολόγησε τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στην κατασκευή και στην εμπορία. Ιδιαίτερα εμένοντας στις περιπτώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. μπορώ να ζητήσω μετά οι συνάδελφοί μου να αναφερθούν στη συγκεκριμένη μελέτη την οποία διαθέσαμε πέρυσι προς το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι όλες αυτές οι σκέψεις και όλα αυτά τα θέματα έχουν πράγματι ληφθεί υπόψη και πεποίθησή μας είναι ότι για να έχουμε μια βιώσιμη αυτοκίνητο βιομηχανία στην Ευρώπη, γιατί είναι ένας βασικός εξαγωγικός παράγων, απαιτείται να υπάρχει ανταγωνιστική αγορά σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο ανταλλακτικών, σε επίπεδο κατασκευής, σε επίπεδο εμπορίας, ακόμα και ε, στο εσωτερικό, αν θέλετε, ε, των ε, επιχειρήσεων εμπορίας αυτοκινήτων που διαθέτουν ένα προϊόν, μία μάρκα, εν πάση περιπτώσει, ένα εργοστάσιο, Θα πρέπει λοιπόν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η βιομηχανία και σε επίπεδο ανάπτυξης και έρευνας και σε επίπεδο διάθεσης τελικού προϊόντος. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι έμποροι και οι κατασκευαστές δεν είναι εχθροί. Μπορεί να έχουν διαφωνίες για το διακανονιστικό καθεστώς, αλλά είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Είτε στη Φιλανδία όπου το multibranding είναι must διότι δεν μπορεί να υπάρξει έμπορος με μία εταιρεία οπότε οι κατασκευαστές δεν διαφωνούν με το multi-branding γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Και στη Γερμανία επίσης όταν υπάρχει υπερβολικό και υπάρχουν προβλήματα μέσω κάθετα ολοκληρωμένων showroom ε, γιατί δεν θέλει η Mercedes σαν παράδειγμα να υπάρχει μια διάχυση της παρουσίας των προϊόντων τους. Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να βρει τους καταλλήλους τρόπους διανομής των προϊόντων τους και αυτό θα πρέπει να το αποφασίζουν φυσικά μαζί οι κατασκευαστές και οι έμποροι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Υφίστανται πιέσεις για την παραγωγή πράσινων αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχουν υπερβολικές διαδικασίες παραγωγής και κάτω από τις συνθήκες αυτές για να διατηρήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και να μην ζητάμε συνέχεια κρατική επιχορήγηση θα πρέπει να βρουν τις πιο ανταγωνιστικές ε, ε, μορφές παραγωγής και πώλησης των προϊόντων τους. Και γι' αυτό στην πρωτογενή αγορά εμείς θέλουμε να εισάγουμε περισσότερο θα έλεγα ευελιξία, περισσότερη ευελιξία. Φυσικά δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τα συνεργεία τα ανεξάρτητα που είναι το άνω του 50%. Όλες αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πολλά πολλές θέσεις εργασίας. Εκεί τίθενται θέματα όπως τα ανταλλακτικά, το είδος των ανταλλακτικών, η πρόσβαση στις τεχνικές ρυθμίσεις και πληροφορίες. Αυτό είναι προς το συμφέρον θα έλεγα και των κατασκευαστών να συνεπάρξουν με αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελπίζω να έδωσα απαντήσεις στις περισσότερες τουλάχιστον από τις ερωτήσεις σας. Mm-hmm. Ίσως κάποιος συνάδελφος για το multi-branding να δώσει περισσότερα στοιχεία. Μα δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Να σας τα πω λοιπόν τηλεγραφικά ότι κάτι δεν συζητήθηκε. Με το ισχύον καθεστώς οι κανόνες του multi δεν χορηγούν την άδεια στους διανομείς να πουλήσουν διάφορες μάρκες. Απλώς δίνουν τη δυνατότητα στην Κομισιόν να εξετάσει περίπτωση την περίπτωση το κατά πόσον θα χορηγηθεί η άδεια αλλά η αλλαγή που προτείνουμε εμείς με το καινούριο σύστημα είναι απριόρι να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην ελευθερία διανομής των κατασκευαστών ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στους καταναλωτές και καταναλώτριες έχει υπολογιστεί στο 20% από την Ισπανική Οργάνωση Διανομέων Αυτοκινήτων. Ανάλογα βέβαια με το κατά πόσον θα είναι εξαιρετική η διαχείριση ή απριόρι καθορισμένη. Γι' αυτό μιλήσαμε για block exemption, για να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες. Όσο για την απασχόληση, υπάρχουν, θα εξισορροπηθούν τα πράγματα μεταξύ των τμήματων της πρότασης. Διότι και οι τέσσερις επιλογές που λάβαμε υπόψη μας δεν προβλέπαν αλλαγή του βασικού συστήματος που δέχονται όλοι, δηλαδή την επιλεκτική διανομή, ποσοτική επιλεκτική, ποσοτικά επιλεκτική διανομή και οι διανομής και οι κατασκευαστές το θέλουν αυτό. Οι διανομής προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από άλλους διανομής. Γι' αυτό υπάρχει το ποσοτικό σύστημα, για να υπάρχει περιορισμένος αριθμός διανομέων. Οι κατασκευαστές συμφωνούν διότι έτσι μπορούν να ελέγχουν τη διανομή του προϊόντος τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του αλλά οι αριθμοί μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε. Οι αριθμοί του περιορισμού δηλαδή. Αυτό θα γίνει και σε περίπτωση αυτή. Άρα δεν υπάρχει αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μήπως οι κατασκευαστές θέλουν να προσθέσουν τίποτα. Πάρα πολύ σύντομα τέθηκαν πολλές ερωτήσεις για τις επιπτώσεις που έχουν οι αλλαγές αυτές στην αηφόρο ανάπτυξη, στην απασχόληση, στα πράσινα αυτοκίνητα κτλ. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μέσα σε μία μελέτη επιπτώσεων όλες τις απαντήσεις. Εγώ μπορώ να σας μεταφέρω την προσωπική μου άποψη. Ο κανονισμός αυτός δεν θα επηρεάσει την παραγωγή των αυτοκινήτων ή την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κτλ για έναν απλό λόγο, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος του. Αν κατασκευάσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα οι κατασκευαστές, οι εταιρείες, οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες θα τα πωλήσουν οι έμποροι. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολύ λίγοι κατασκευαστές που έχουν μεγάλα κέρδη σε αυτή τη φάση και πολύ λιγότεροι έμποροι που σε αυτή τη φάση κερδίζουν χρήματα. Είμαστε σε ένα τομέα ο οποίος δεν δίδει πάρα πολύ ψηλά κέρδη και πριν την κρίση πολλοί εμποροί δεν κέρδισαν πολλά χρήματα και κάτι πρέπει να κάνουμε από κοινού. Αν κλείσουν τα επόμενα χρόνια κάποιοι έμποροι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τον κανονισμό εξαίρεσης, αλλά με το ότι δεν υπάρχει ζήτηση για να πωλήσουν αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας. Τώρα γιατί πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή είναι μια καλή πρόταση. Αυτό το κάνουμε γιατί εν πολύ αναιρεί κάποιους από τους περιορισμούς που είχαμε σε σχέση με τον κανονισμό αυτό. Αν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν μεγαλύτερο θα έλεγα ρόλο να παίξουν και στη δημιουργία των δικτύων εμπόρων, αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει γενικότερα. Τα δίκτυα των εμπόρων πιέζονται αυτή τη στιγμή, πιέζονται πάρα πολύ και μαζί με τους κατασκευαστές θα προσπαθήσουν να βγουν τις κατάλληλες λύσεις και δεν είναι σωστή ιδέα να αφήσει κανείς την έβρεση των λύσεων αυτών στους επίσημους εμπόρους. Ναι. Βρίσκουν κάποιες λύσεις οι οποίες είναι καλές για αυτούς αλλά όχι για όλους. Ναι. Και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να έχουμε δίκτυα που να εξυπηρετούν τους πολίτες, τους καταναλωτές. Δεν στέλνουμε εμείς επιστολές τερματισμού συνεργασίας στους εμπόρους, εμείς θέλουμε να έχουμε σωστή συνεργασία με εμπόρους οι οποίοι να πηγαίνουν καλά οικονομικά και να είναι χρήσιμοι για τους αγοραστές. Ένα τελευταίο σημείο <clears throat> για μια χώρα σαν τη Φιλανδία. Σε επίπεδο multi-branding, σας το είπα και πριν, στη Φιλανδία τυπικά υπήρχε multi-branding και πριν εμείς προχωρήσουμε στον κανονισμό εξαίρεσης. Υπήρχε multi-branding κατά τη διάρκεια όλων των ρυθμίσεων που ίσχυσαν τα τελευταία χρόνια και μπορεί να πιστεύει κανείς λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της χώρας ότι θα συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το multi-branding στο μέλλον γιατί οι κατασκευαστές δεν έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να διαθέτουν αποκλειστικά δίκτυα σε μια χώρα σαν τη Φιλανδία και αυτό ισχύει για όλη τη Σκανδιναβία μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Μια γενική παρατήρηση από πλευρά των εμπόρων. Είναι προς το συμφέρον των κατασκευαστών, των εμπόρων και των υπαλλήλων και των καταναλωτών να διαθέτουν η δίκτυα, θα έλεγα, επιλεκτικής διανομής για να δώσουμε τη σημασία και την ποιότητα στο προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν το δίκτυο των εμπόρων να μπορεί να καλύπτει και να είναι σε θέση να αποσβέσει τις επενδύσεις τις οποίες κάνει παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες των καταναλωτή. Ο προτινόμενος κανονισμός στην ουσία θα δημιουργήσει μια ρήξη στην ισορροπία την ευαίσθητη που υπάρχει σήμερα στη σχέση ανάμεσα σε εμπόρους και κατασκευαστές και ο κανονισμός αγνοεί τις μαζικές επιδοτήσεις οι οποίες υπάρχουν στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, ανάμεσα δηλαδή στο aftermarket και την πρωτογενή αγορά. Η πρωτογενής αγορά σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ πιεσμένη όπως ξέρετε και τα περιθώρια κέρδους είναι ελαχιστότατα. και νομίζω το να πούμε ότι μόνο οι κατασκευαστές θα αποφασίσουν το εύρος και το μέγεθος των δικτύων διανομής, αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα, θα οδηγήσει σε κλεισίματα επιχειρήσεων και θα υποστούν οι πρωταγωνιστές της αγοράς αυτής και σε επίπεδο πρωτογενούς αγοράς και σε επίπεδο aftermarket απαράδεκτες πιέσεις και ο ανταγωνισμός ο οποίος έχει έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί σήμερα δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί στο τέλος και αυτό φυσικά θα ευνοήσει χώρες εκτός Ευρώπης, χώρες επίσης οι οποίες αναπτύσσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν πάρα πολλές δυσκολίες να τα διανύμουν αν δεν υπάρχει ε, multi-branding εκτός βέβαια και αν δώσει τις ευλογίες του κατασκευαστή. Ευχαριστώ. Ήθελα να επανέλθω στο Monte μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ όμω πρέπει, θέλω να σου πω ότι πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μια κοινή αγορά και θα πρέπει οι καταναλωτέ να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν διαφορετικών μάρκων αυτοκίνητων χωρί να πρέπει να τρέχουν πάνω κάτω. Η Ευρωπαϊκή Ώρα δίνει λιγότερε επιλογέ και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Δεν ε, αρκεί να βασιζόμαστε σε εθελοντικέ συμφωνίε γιατί είδαμε στο παρελθόν ότι κάτι τέτοιο δεν οδηγεί στο στόχο του. Όσον αφορά τη λεγόμενη αγορά κατόπιν πώληση στο του. υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Θέλω να πω σε εκείνου που ανησυχούν για την απασχόληση ότι αυτή η αγορά προσφέρει τοπικέ ε, θέσει απασχόληση που δεν μπορούν να μεταφερθούν λίγορα κάπου αλλού γιατί είναι οπωσδήποτε σταθερέ στην περιφέρειά σα στις χώρε σα, Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόβλημα και θα ήθελα να εθαρρύνω όλου να λάβω υπόψη όλε τι αλλαγέ του τομέα. Γιατί συμφωνούμε ότι οι κατασκευαστέ των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν προβλήματα, υπάρχει όμω μια ολόκληρη αλυσίδα που παίζει ένα σημαντικό ρόλο και για το καταναλωτή αλλά και για την απασχόληση. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας πω ότι η FIA θα ήθελα να διασφαλίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών για αυστηρή, ε, καθαρή και πράσινη κινητικότητα. Και ελπίζω ότι οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτος. Και να σε μια πιο γενική ε, απάντηση γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί το BR αυτή τη στιγμή. Έχω να σας πω χρειαζόταν να αλλάξει η νομοθεσία αυτή λόγω των αυξανωμένων δυσκολιών που προκαλούνται από τη χρήση υπολογιστών στα αυτοκίνητα. Οι κανόνες οι σημερινοί δεν καλύπτουν λοιπόν όλα τα προβλήματα των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά θέματα εγγύησης. Τελειώνοντας έχω να πω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πλήρη ορισμό του τι είναι τεχνική πληροφορία στο επόμενο mini BR και την δυνατότητα να εξασφαλιστεί και να διασφαλιστεί το multi-branding. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μάκαμες μου ζήτησε να πει δύο λόγια και θα του δώσω το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία εδώ, δεν έχουμε όμως πάρα πολύ χρόνο. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια για το ψήφισμα που προετοιμάζει η Επιτροπή σας που οπωσδήποτε θα συμβάλλει. Αν μου επιτρέπετε να στραφώ στην κατεύθυνση που έχει η συζήτηση, θα συμφωνείτε ότι καλύφθηκε σε γενικές γραμμές όλα τα δομέα, αλλά κάτι που πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι το εξής. Η Κομισιόν είπε ότι οι κατασκευαστές θέλουν η ευελιξία να μεταφερθεί στους, στις αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων. Την άλλη μεριά οι αντιπροσωπείες, οι έμποροι δηλαδή, λένε ότι εντάξει θέλουμε περισσότερη ευελιξία, η ευελιξία όμως αυτή δεν θα οδηγήσει σε αρκετή δυνατότητα ευελιξία σε εμάς για να κάνουμε στις επιχειρήσεις μας. Αυτό ήταν όμως ε, ο στόχος της πρώτης 2002. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο η Κομισιόν όταν έκανε την αξιολόγηση των επιπτώσεων που διάβασα είναι πάρα πολύ πιστική για το γεγονός ότι η επανεξορρόπηση της ε, ευελιξίας θα μπορέσει να προσφέρει γενικά εξισορρόπηση των ε, δημοσιογράφων και των συμφερόντων καταναλωτών. Δεν είμαι λοιπόν φεβισμένος ότι αυτές οι πτυχές των δυνατότητων των καταναλωτών έχουν ληφθεί υπόψη. Επίσης η Κομισιόν τόνισε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα της ε, δυνατότητας επιβολής των νησιών των κανόνων. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι οι καινούργιοι κανόνες αποτελούν σημαντική πρόοδο. Λοιπόν, εάν η επιβολή είναι το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, οι αλλαγέ που γίνονται δεν νομίζω ότι μας προχωρούν. Ομολογώ λοιπόν, εγώ έχω ασχοληθεί εδώ και ένα χρόνο με το θέμα αυτό και έχω πάντα τονίσει το θέμα της ανάγκης αλλαγών. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα επιχειρήματα έχουν αποδειχθεί πιστικά. σημειώνω αυτό που είπαν οι ε, έμποροι όσον αφορά το 30%. Όταν εγώ πριν από μερικά χρόνια έκανα μια έρευνα εδώ, προσπαθήσα να αποδείξω ότι το κόστος που αναφερόταν ήταν πολύ ψηλό, γιατί το πραγματικό κόστος λόγω των εκπτώσεων που δίνονται από τους εμπόρους και τις αντιπροσωπείες και λοιπά ήταν πολύ χαμηλότερο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Παραμένει όμως ε, αληθές κύριε Πρόεδρε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό που είναι. Χρειαζόμαστε όμως κάποια σταθερότητα που κατά γνώμη θα μπορούσε να επιτευχθεί συνεχίζοντας τη σημερινή κατάσταση μερικά χρόνια. Έχουμε όμως την πρόταση μπροστά μας, πρέπει να τη σεβαστούμε και η Κομισιόν είναι εκείνη η οποία έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και το δικαίωμα εκτέλεσης στον τομέα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα στα πλαίσια του δικού σα ψηφίσματο θα μπορέσουμε να τονίσουμε κάποια σημεία, ακόμα και αν η Κομισιόν είναι τελευταία λύση αγνόηση. Θα πρέπει να δούμε όμω ποιε είναι οι επιπτώσει κατόπιν. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάλκομ. Είναι πολύ σαφέ νομίζω. Πολύ φοβούμαι ότι τελικά θα έχουμε αφήσει τα πράγματα ημιτελή. Υπάρχει μια πρόταση προφορικής ερώτησης και μια πρόταση ψηφίσματος που έχει ε, μοιραστεί. 14 Απριλίου είναι η προθεσμία για σχόλια από αυτόν και θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε από αυτόν στην συνεδρίασή μας της 19ης Απριλίου. Mm -mm. Παρακαλώ λοιπόν το γρηγορότερο δυνατόν τα σχόλιά σας στη γραμματεία. και θα προσπαθήσουμε να οργανωθούμε κατά δυνατόν καλύτερα μέσα στα πλαίσια αυτών των πολύ στενών προθεσμιών. Και ο στόχο μα είναι να ψηφίσουμε στην πρώτη σύνοδο ολομιλίας του Μαΐου. Μαΐου. Για να έχουμε απόλυτα τοποθετηθεί πριν να πραγματοποιηθούν οποιασδήποτε αλλαγέ του κανονισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν στην συζήτησή μας και που συνέβαλαν σε αυτή και άλλοι συνέβαλαν σημαντικά και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι διαβάζουν τις συμβολές που υποβάλλονται για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε παρόντος. Σε λίγα λεπτά θα προχωρήσουμε στους μία πέντε σημερισίες διάταξεις. Ευχαριστώ. Right, we will Καλώς σας ευχαριστώ. Περνάω τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Γι' αυτό όσοι θέλετε να συνεχίσετε ιδιωτικές συζητήσεις εκτός εθούσης. Εκτός Δεν μπορεί ο εισηγητής να σας υφίσταται. Ακούσατε τι είπα για την ακρόαση που θα κάνουμε την Τετάρτη που απόγευμα σχετικά με τα μαθήματα που πήραμε από το ελληνικό παράδειγμα. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να περιοριστούν σε ένα θέμα, όχι πολυμερείς ερωτήσεις ή πολυθεματικές ερωτήσεις και θα πρέπει να ε, εκφέρονται μέσα σε ένα λεπτό. Καλό θα ήταν επίσης να υπάρξει και μία σύντομη συζήτηση με τους υπαλλήλου και τους συντονιστές που θα μείνουν εδώ μετά από αυτή τη συνάντηση. Δεν είναι μία επίσημη συνάντηση συντονιστών. Απλά θα έλεγα είναι μία προσπάθεια ενημέρωσης για καλύτερη συστηματοποίηση των ερωτήσεών μας. Περνάμε τώρα στην διασυνοριακή διαχείριση της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Συντονίστρια είναι, η συγγήτρια μάλλον, η κυρία Φερέρα. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία και δίνω το λόγο αμέσως στην Ελίσσα. Θα μιλήσω αγγλικά, λέει η Ελίσσα, για να πάνε πιο εύκολα τα πράγματα. Μετά την πρώτη μου βάψεων για την έκθεση αυτή που έλαβε χώρα στις 22 του μηνός, εργαστήκαμε σκληρά στην ε, παγίωση των απόψεών μας. Στην αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εκτελεστική Επιτροπή, του εκπροσώπου βιομηχανία, εκκρεμονιστέ, επιτηρητέ, επιθεωρητέ, ε, πολιτικού, ακαδημαϊκού κύκλου και του κοιόδε εισηγητέ για τον ανοιχτό πνεύμα και τις συμβολές τους μέχρι στιγμής. Και αποτέλεσμα θα συνεχίσουν ναι, με το ίδιο πνεύμα. Θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως τη γραμματεία για την βοήθεια που μου προσέφερε, τη γραμματεία της ΕΚΟΝ ιδίως. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω την πολύ σημαντική μας ακρόση της 16 Μαρτίου τη διάσκεψη των Κομισιών στις 19 Μαρτίου και επίσης μια ειδική διάσκεψη που οργάνωσε στις 26 Μαρτίου στη Λισαβόνα. Μέσα όλων αυτών είναι πολύ καθυσιστικό και ενδιαφέρον να καταλάβουμε ότι υπάρχει συνένεση σε υψηλό επίπεδο παρόλες τις δυσκολίες του θέματος. Συνένεση αυτή όμως δημιουργείται λόγω της ανάγκης της, ε, του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεμπεσόπιση κρίσεων αυτού του τύπου και τις γενικές κατευθυντικές γραμμές. Μεταξύ όλων αυτών των σημαντικών θεμάτων θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι υπάρχει μια πεποίθηση των εμβαλωμένων ότι θα πρέπει να δούμε τριπλά αυτό το θέμα, δηλαδή να επανεθέσουμε και να εξετάσουμε τη νέα δομή εποπτείας κατόπιν να ενδυναμώσουμε τους κανονισμούς όσον αφορά το κεφάλαιο και τρίτον τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δυνατότητας ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων. Οι εργασίε γίνονται και στα τρία αυτά μέτωπα και το Κοινοβούλιο έχει οπωσδήποτε ιστορικό ρόλο να παίξει για να τα πετύχουν ε, τα πράγματα αυτά όπως πρέπει. Η έκθεση αυτή ελπίζω θα συμβάλλει προς αυτό το πνεύμα συνοχής. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ρεαλιστική αλλά φιλόδοξη πρόταση που θα πετύχει ευρεία συνένεση μεταξύ όλων. Αυτό είναι το πνεύμα βάσει το οποίο εργαζόμαστε. Επειδή έχουμε τώρα την έκθεση, το σχέδιο έκθεση μπροστά μας, δεν θέλω να επισέλθω στις λεπτομέρειες, αλλά να τονίσω τις κύριες τέσσερις συστάσεις. Πρώτον, ε, ε, θέτουμε φιλόδοξους στόχους για να πετύχουμε τελικά μια, ένα κοινό ψήφισμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πράγμα το θέμα, θα είναι πολύ χρονοβόρο, αλλά μεταξύ υποστηρίζουμε μία μέθοδο εκ των κάτω προς τον άνω. Και τη δημιουργία ενός πλαισίου ευρωπαϊκού. Αυτό τι σημαίνει, θα πρέπει να ακούμε τους, την ομάδα των επιθεωρητών, θα πρέπει να φροντίσουμε πάντα τους εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών βάση πάντα της δομής του Μνημονίου Συνεννόησης που καταρτίστηκε το 2008. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται ε, υπό την αιγίδα της νέας αρχής ΕΜΠΑΝ. Αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα καθορίζει ένα νέο κοινό ε, ένα νέο κοινό σύνολο κανόνων, της ε, διατάξης που αφορούν τις πτωχές της, Τρίτο, να δούμε, να ξέρουμε το πώς θα αντιδράσουμε αν υπάρξει κρίση. Και επίσης, ποια θα είναι η πραγματική αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης. Ε, θα πρέπει να έχουμε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε στενή συνεργασία με τις ομάδες εθνικών επιθεωρητών και τις ομάδες σταθερότητα για τις, τη μη συστηματική προσέγγιση θα πρέπει να βρισκόμαστε πάντα μέσα στα πλαίσια του δομισμού της ΕΜΠΑ και στην εργασία με τις ομάδες σταθερότητας διασυνολικής αντιμετώπισης κρίσης. Η παρέμβαση αυτών των επιθεωρητών και εποπτών θα πρέπει να βασίζεται σε σημαντικά ε, μέσα και θα πρέπει να ναι. υπάρχει ένα σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια αξιολόγηση εποπτείας που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός σταθερού διαφανούς μηχανισμού βάσει του οποίου θα αποφασίζεται η παρέμβαση ή μη. Κλάδι. Εκτός από αυτά, θα πρέπει να εργαστούμε για να έχουμε στα χέρια μας τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν αυτοί οι υπόπτες να παρεμβαίνουν όπως πρέπει και όποτε πρέπει. Είναι μακρά η απόσταση που πρέπει να διανύσουμε μέχρι το... εκεί. Τα Risk τα στην πρώτη φάση θα έχουμε μια μικρή ομάδα των λεγόμενων θεσμικών πιστοτικών οργάνων που αποτελούν το 70% του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ίσως μπορούμε να φτάσουμε μόνο στο ύψος 40-50%. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά για να μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Στην πρώτη φάση. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά τα θεσμικά πιστοτικά ιδρύματα και αυτή είναι η δεύτερη σύσταση. Για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι που να μπορούμε να αποκαλέσουμε ευρωπαϊκό νόμο επιχειρήσεων τραπεζών, όπως τον ευρωπαϊκό νόμο επιχειρήσεων, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί υποχρεωτικά από όλα τα θεσμικά πιστοτικά ιδρύματα. η εποπτεία των συστημάτων θα είναι ένα δεύτερο στοιχείο για το ειδικό αυτό καθεστώς των θεσμικών ε, πιστοτικών ιδρυμάτων. Η ΕΜΠΑ θα μπορεί να παρεμβαίνει σε ορισμένα επίπεδα όταν έχει φτάσει το σημείο εκκίνησης των μέτρων και το Συμβούλιο Αντιμετώπισης του Κινδύνου θα πρέπει να ορίσει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μία τράπεζα θεωρείται θεσμικό πιστοτικό ίδρυμα και να προτείνει ταυτόχρονα καταλόγους δημοσίους αυτών των ιδρυμάτων που θα πρέπει να κρατούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κινδύνου Συστομικών ε, Πιστοτικών θεσμικών συγγνώμη πιστοτικών ιδρυμάτων. Μετά, τι το θέμα της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων. Γιατί δεν χρησιμεύει να υπάρχουν οι δυνατότητες παρέμβασης χωρίς να υπάρχουν οι πόροι παρέμβασης. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο σταθερότητας που θα ε, τη χάνει δημόσια ε, αλλά και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός ταμείου και όχι ενός ε, επιδόματος γιατί αυτό θα είναι πιο σαφές, θα είναι πιο εύκολο να παρέμβει και θα ενδυναμώσουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της διαχείρισης της αποτυχίας. Αυτό θα είναι απογορισμένο από τη Γενική Διεύθυνση ΕΣΥΣ, που έχει άλλο ρόλο να παίξει. That would make these funds αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο και το ταμείο αυτό θα πρέπει να τη χάνει διαχείρισης βάση κατευθυνίων γραμμών που θα τονίζουν την ασφάλεια, την ρευστότητα και θα ακολουθούνται επίσης οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι. Θα χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί εφόσον ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο που να διατίθεται η ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Έχουμε κάθε συμφέρον και αυτή ήταν και η απόφασή μας να αποφύγουμε συμπληρωματικό κόστος και υπερβολική γραφειοκρατία. Και γι' αυτό η ενίσχυση τεχνικής μορφής της διαχείρισης του τομείου θα πρέπει να γίνει όχι με μια νέα υπηρεσία, αλλά να γίνεται από τα πλαίσια των τραπεζικών αρχών. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια μονάδα η οποία θα μπορούσε αν χρειαστεί σε περίοδους κρίσης να ενισχύεται από τους εθνικούς επόπτες αυτή τη στιγμή όμως δεν προτείνουμε να δημιουργηθεί περισσότερη γραφεία και περισσότερη πολυπλοκότητα και κόστος στο σύστημα. Τελικά, έχω να παρατηρήσω ότι θα πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα τσουνάμι νέων κανονισμών και απαιτήσεων. Είναι αληθές ότι αυτή είναι μία από τις πτυχές που έχουμε πάντα κατά νου. Από την άλλη μεριά όμως επίσης αληθές ότι τώρα και εδώ πρέπει να δράσουμε. Θα πρέπει δηλαδή οι προτάσεις του Κοινοβουλίου να είναι φιλόδοξες, ταυτόχρονα όμως λογικές και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. Αυτές οι πτυχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο να εξετάζουμε τις συμβολές σε ένα ταμείο σταθερότητας που θα πρέπει να υπολογιστούν σε μακρά χρονικά διαστήματα. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει οι συμβολές στο ταμείο αυτό να συμβάνουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα θεσμικά πιστοτικά ιδρύματα. Και αυτή η πρόταση βέβαια θα απαιτεί συμπληρωματικούς ορισμούς και διαβουλεύσεις με τις βασικές επιτροπές. Γνωρίζουμε επίσης πλήρως ότι η επιλογή για τη γλίγορη παρέμβαση των θεσμικών ε, αυτών πιστοτικών ιδρυμάτων θέτει κάποια προβλήματα, δηλαδή η προσέγγιση σε δύο επίπεδα, ανάλογα τα πόσο ένα ίδρυμα θεωρείται ε, θεσμικό ή όχι. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ανάμεσα όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ένα επίπεδο πεδίο παιδιάς Αλλά αυτό που προτείνεται εδώ είναι ένα πρώτο βήμα για προοδευτική δημιουργία ενός πιο ευρωπαϊκού πλαισίου. Αυτό μου φαίνεται λογικό. Και τέλος, για να είμαστε αποτελεσματικοί, όσον αφορά την ε, πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, απαιτείται συνοχή. Η συνοχή είναι σημαντική μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών που υπάρχουν, ιδίως αυτή εδώ της έκθεσης και του ρόλου που αποδίδει το Κοινοβούλιο στις αρχές και προφανώς θα τονίσω και την έκθεση των ε, τραπεζικών αρχών που προτιμάζει ο συνάδελφος Καρθία Μαργάλιο και την γενική οδηγία του ΖΕΣ προσέτο. Αυτά όλα θα πρέπει να ενδυναμωθούν, να συντονιστούν, ούτω ώστε η θέση του Κοινοβουλίου να είναι συνοπτική, συνεκτική Μέχρι στιγμής βλέπω ότι μπορούσαμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, ιδίω όσον αφορά αυτό το Ταμείο Σταθερότητας που χρηματοδοτείται από τις ε, ε, λόγω οικονομικούς κύκλους. Λοιπόν, εγώ βασίζομαι στη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους για να μπορέσει η παρούσα πρόταση να πετύχει τον απότερο στόχο μας, να δυναμώσει δηλαδή τη σταθερότητα, την ισχύ και την εθνική αναγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστικού συστήματος, ταυτόχρονα βασιζόμενοι στα μαθήματα του παρελθόντος και εξασφαλίζοντας και προστασεύοντας όλους τους αματιαμευτές και τους φορολογούμενους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την προσοχή σας, για το ενδιαφέρον σας και βασίζομαι στις συμβολές σας για το μελόν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Elisa. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δω πού είναι ο κατάλογος λοιπόν. Η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσουν συγχαίροντας την Ελίσα για την έκθεσή της είναι φιλόδοξη και υποστηρίζω τις περισσότερες από τις συστάσεις της προς την Κομισιόν. Υπάρχουν όμως μερικά θέματα που θέλω να θίξω, θέματα δηλαδή είτε που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση είτε που νομίζω ότι θα ήταν σημαντικά για να πετύχουν τα προτινόμενα μέτρα ή συστάσεις λόγω της κρίσης. Πρώτον, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε καλύτερα το θέμα των εμβασμάτων μεταξύ της ίδιας χρηματοπιστωτικής, του, ίδιου χρηματοπιστωτικού ομίλου, μέσα στον ίδιο χρηματοπιστωτικό όμιλο και το έμβασμα είναι ένας τρόπος μεταφοράς βέβαια ρευστότητας από μια θηγατρική προς το κέντρο συνήθως. Οι πιστωτέ νομίζω ότι καταλήγουν πολλές φορέ επειδή δεν υπάρχει αυτό το ενιαίο σύστημα εμβασμάτων, να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, όπως λέει και η σύσταση 1-1. Ότι δηλαδή ο στόχος είναι να ενισχυθεί η θέση των καταθετών και να υπάρξει εγγύηση ίσης μεταχείρισης τους μεταξύ διαφόρων χωρών. Στην πρόταση αναγνωρίζεται η ανάγκη να υπάρξει ένα, μια καλύτερη διευθέτηση του θέματος του κόστους όλων αυτών των τραπεζικών λειτουργιών. για να υπάρχει η απαραίτητη ρευστότητα που να χορηγείται και στις θηγατρικές όποτε το ζητήσουν οι πελάτες τους. Τώρα για τις διαμεθοριακές τράπεζες και την περίπτωση πτωχεύσεων είναι προφανές ότι καλύτερα είναι το θέμα αυτό να λυθεί ενωσιακά είτε μέσω εναρμόνισης που από ό,τι καταλαβαίνω είναι και η άποψη της συντάκτριας, είτε μέσω ενός ενιαίου ενωσιακού καθεστώτος όπου ο τραπεζικός όμιλος θα θεωρείται ένα ενιαίο σύνολο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερο όμως σχόλιο, ο διαχωρισμός που προτείνεται στην έκθεση μεταξύ θεσμικών και μη θεσμικών διαμεθοριακών τραπεζών. Αναλύοντας τα υπέρ και τα κατά κατέληξα ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός θα δημιουργήσει μάλλον περισσότερα προβλήματα από ότι λύσεις. Ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε ποσοτικά κριτήρια για να καθορίσουμε ποιες τράπεζες είναι θεσμικές και ποιες δεν είναι. Τελικά θα είναι αυθαίρετη η διαδικασία και το αποτέλεσμα. Και τέλος όπως έδειξε και η τελευταία κρίση οι τράπεζες που θεωρούνται μη θεσμικές τελικά καταλήγουν να γίνονται θεσμικές και να χρειάζονται βοήθεια από τα κράτη παρόλα αυτά. Απ' την άλλη, το να χορηγηθεί η ετικέτα θεσμική σε περιορισμένο αριθμό τραπεζών θα σήμαινε κατά κάποιον τρόπο ότι είναι κεντρικές ως προς τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ότι μόνο αυτές ή κατά κύριο λόγο αυτές πρέπει να σωθούν σε περίπτωση προβλήματος. Άρα στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός με άλλες τράπεζες. Γι' αυτό νομίζω ότι πιο λογικό θα ήταν να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς σε, όλες τις, σε όλους τους διαμεθοριακούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους με όλες τους συστηγατρικές. Η κρίση μας έδειξε ότι πράγματι υπάρχει αυτή η τάση να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης ορισμένες κεντρικές τράπεζες αντί ορισμένων άλλων τοπικότερων ενώ εμείς θέλουμε ίση μεταχείριση των καταθετών και των πιστωτών των. Και από αυτό βγαίνει και το συμπέρασμα ότι το κολέγιο των εποπτών πρέπει να είναι ενεργό καθ' τη διαχείριση μιας κρίσης, εθνικά και διαμεθοριακά. Άρα όλες οι διαμεθοριακές τράπεζες, θεσμικές ή μήνα έχουν την ίδια μεταχείριση. Και τέλος τέλος, τώρα που εξετάζουμε το μέλλον, θα έπρεπε να δούμε μήπως δεν θα ήταν χρήσιμο επίσης να δούμε και πώς λειτουργούσαν οι τράπεζες πριν αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα που κατέληξαν στην κρίση. Μια τελευταία έκθεση από τον ΟΣΑ είναι σχετικός πολύ ενδιαφέρουσα γιατί ο ΣΑ προτείνει μια επιστροφή στο παλαιότερο σύστημα, δηλαδή από το γενικευμένο τραπεζικό σύστημα σε, στο παλαιότερο σύστημα μιας τραπέζης holding. Μπορεί κανείς να πει πολλά υπέρ και κατά του συστήματος αυτού, αλλά ένα τέτοιο πρότυπο θα σήμαινε ότι όλες οι τραπεζικές λειτουργίες επιτρέπονται, αλλά τα κέρδη των τραπεζών συγκεφαλαιώνονται γενικά. Και όσο για τα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης κρίσεων, θα μπορούσαν οι τράπεζες να τα εφαρμόσουν ανεξάρτητα από τη γενικότερη λειτουργία τους αλλά τελικά τα προβλήματα σε έναν τομέα λειτουργίας μιας τράπεζας δεν θα καταλήγουν αναγκαστικά να έχουν επιπτώσεις και στους άλλους τομείς της λειτουργίας της. Δεν ξέρω κατά πόσον η πρόταση αυτή του ΩΣΑ είναι σοβαρή και ρεαλιστική, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Και τρίτο τέλος της ομιλίας μου, ως σκιώδης θα ήθελα να πω ότι συνεργάστηκα πολύ καλά με την Ελίσσα και νομίζω ότι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον έγκυνται στο να δημιουργηθεί ένα σύστημα καλύτερης διαχείρισης των κρίσεων που να μην όμως ζημιώσει τη λειτουργία των τραπεζών και σε κανονικές περιόδους λειτουργίας χωρίς κρίση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από τις ε, παρατηρήσεις της κυρία Σουίμπερ, λέει η κυρία Σουίμπερ της ε, κυρία Χούμπνερ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ και την κυρία Φερέιρα για την τεράστια προσπάθεια που έκανε κατανοώ αυτά που είπε ότι το σύστημα δουλεύει καλά για τις μικρές και τις μεσαίες τράπεζες και ο εναρμονισμός ε, σε ένα πρώτο επίπεδο ε, των, κριτηρίων για την αξιολόγηση της ρευστότητας κτλ. είναι κάτι που ακούγεται εύκολο αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί εύκολα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με επιστοτικά ειδήματα σε διαφορετικές χώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω σαν παράδειγμα πως ε, η υπεύθυνη αρχή, ε, η ευρωπαϊκή, θα είναι αρκετά ισχυρή και μεγάλη σε επίπεδο προσωπικού για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αν καταλαβαίνω καλά, κάποιες από τις ε, μεγάλες τράπεζες στην τελευταία κρίση υπήρχαν 60 εκπρόσωποι της ρυθμιστικής αρχής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ θα πετηθούν εφόσον θέλουν να λειτουργήσουν συνολικά καλά ε, τεράστιοι αριθμοί υπαλλήλων. Όταν υπάρχει δηλαδή μια σφαιρική τράπεζα, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με τους ε, παγκόσμιους ρυθμιστές όταν έχουμε να κάνουμε με Αμερικανούς, Ασιάτες κτλ ιδιαίτερα όταν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πτώχευσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υπάρχει πολύ σημαντική έκθεση και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις άλλες αγορές ε, υπάρχει πρόβλημα. Η λογική πολύ μεγάλη για να σωθεί ή πολύ μεγάλη για να αποτύχει μια τράπεζα είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σώσει την τράπεζα αυτή όσο μεγάλη και να είναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλες προτάσεις και άλλα μέτρα. Έγινε μια πρόταση από τον Πολ Τάκερ ότι μια δυνατότητα η οποία ελέγχει τα επίπεδα των swaps να συμβαίνει νωρίτερα όπως επίσης να υπάρχουν και εσωτερικά στοιχεία πληροφόρησης για τα κεφάλαια της τράπεζας. Οι τράπεζες επίσης θα πρέπει να εκδίδουν ομόλογα δεκαετή τα οποία να αντιστοιχούν με το 10% του χρέους τους. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέπει να κατανοούμε καλύτερα ε, τους ε, λογαριασμούς αυτών των τραπεζών και να αναλαμβάνουν μόνες τους τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και όχι τόσο να περιμένουν από τον φορολογούμενο. Πώς όμως θα πιέσουμε μια μεγάλη τράπεζα να πάρει μέρος σε ε, ένα τέτοιο σχήμα θα έλεγα και να μην μετακινηθεί απλά σε μια άλλη νομική δικαιοδοσία, να πάει δηλαδή σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Οι μηχανισμοί μας <clears throat> δεν μπορούν να απαγορεύσουν την εισρωή κεφαλαίων από ένα πιστοτικό ίδρυμα στην μητρική εταιρεία. Είδαμε τι έγινε με την εταιρεία Lehman Brothers. Δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε την κίνηση των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τα χρήματα μάλλον από συνταξιοδοτικά ταμεία να μετακινούνται εκτός Ευρώπης λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης του πιστοτικού ιδρύματος. Δεν μπορούμε λοιπόν έστω και εν μέρη να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των πολύ μεγάλων θα έλεγα πιστοτικών ιδρυμάτων. Αλλά βέβαια για τις μεσαίες επιχειρήσεις, τις τραπεζικές, ε, το σύστημα αυτό έτσι όπως προτείνεται μπορεί να είναι ευεργετικό. Σβέν. Και εγώ θα ήθελα... Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίσσα για την εξαιρετική της εργασία με την οποία συμφωνώ, τουλάχιστον με τα περισσότερα από όσα λέει η έκθεσή της και τη βασική της γραμμή. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ορισμένα από τα σωστά θέματα που έθιξε, όπως τα θέματα της έδρας και των θυγατρικών ή τα προβλήματα του ορισμού του τι είναι θεσμικό θεσμικός και τι δεν είναι θεσμικός όμιλος. Όλα αυτά πολύ καλά τα εξέφρασε, αν και χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Γι' αυτό θα περιοριστώ σε τρία πρόσθετα θέματα, επί των οποίων θα ήθελα να συνεχίσω να συνεργάζομαι με την Ελίσσα και τους άλλους κοιόδης. Πρώτον, στην έκθεση δεν είναι σαφές ότι θα θέλαμε οι πιστωτές να πληρώνουν πολύ περισσότερο τμήμα του βάρους ε, της στήριξης ε, προβληματικών επιχειρήσεων από ό,τι μέχρι τώρα. Δεν το, το λέει μεν, αλλά όχι πολύ σαφώς. Σε τι βαθμό δηλαδή πρέπει οι πιστωτές να θεωρούνται υπεύθυνοι για τις αποτυχίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν αρχίσουν οι αποζημιώσεις και οι στηρίξεις. Έπειτα, αναφέρατε την πρόταση του ΟΣΑ και του θέματος του περιορισμού των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Στην πρόσφατη κρίση όμως δεν είδαμε απλώς τον κίνδυνο του να υπάρχουν μεγάλες τράπεζες που θεωρούσαμε ότι ήταν αδύνατο να αποτύχουν, αλλά και την υπερβολική αύξηση των δραστηριοτήτων τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μέγεθος θα θέλαμε να έχουν οι τράπεζες και άρα πώς το σύστημα αυτό, το νέο καθεστώς διαχείρισης τέτοιων κρίσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενθάρρυνση δημιουργίας μικρότερων τραπεζών μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας μάλλον παρά τεραστίων ε, θεσμικών ή μη θεσμικών και πολιτικά σημαντικών τραπεζών. Αυτό το θέμα του μεγέθους λοιπόν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επανέλθουμε όταν θα συζητήσουμε το θέμα της μεταρρύθμισης ε, when we talk about... Ε, του cd 4 και της λειτουργίας του προτινόμενου ταμείου. Τέλος, υπάρχει και το θέμα σε ποιο βαθμό η πολιτική του ανταγωνισμού δεν θα μπορούσε να παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο από ό,τι μέχρι σήμερα. και τις σχέσεις μας ως προς αυτό με τους Αμερικανούς. Υπάρχει πρόταση Βόλκερ που ανταποκρίνεται αρκετά σε αυτά που συζητάμε και εμείς εδώ. Τέλος, μόνον οι θεσμικές τράπεζες διατρέχουν κίνδυνο ή μήπως θα μπορούσαν και τεράστια ταμεία που δεν είναι τράπεζες να θεωρηθούν ανάλογα επικίνδυνα. Υπάρχει η έκθεση ΕΣΜΑ που θέτει το θέμα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν τράπεζα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς συνδέονται τα θέματα των τραπεζών με τα θέματα των ταμείων. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω, προσδοκώ στις, ε, τις επόμενες συζητήσεις. Μάλιστα σας ευχαριστούμε. Θα σας διαβάσω ποιοι θέλουν να ζητήσουν το λόγο για να δείτε αν θέλει κανείς να προσθεθεί. Ford, Astrid Lulling, Pavanche Beres, Peter Skinner, Antolin Sanchez Prezado, Jürgen Klut and myself. Any, anybody else? Κανείς άλλος, καμία άλλη? Όχι, εντάξει. Ωραία. τεφίκη. Οι ερωτήσει μου είναι για το τι μπορεί να κάνει κανείς πριν από την πτώχευση ενός πιστοτικού ιδρύματος έτσι ώστε να αποτραπεί αν θέλετε η δυνατότητα αυτή. και να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε τον τελευταίο καιρό. Για το πρώτο σημείο της εισηγήτριας βάζει πάρα πολύ καλούς στόχους. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τους στόχους. Γιατί χρειαζόμαστε τον τομέα αυτό, γιατί χρειαζόμαστε πρόσβαση στο κεφάλαιο και χρειαζόμαστε επίσης να ελαττώσουμε τους κινδύνους τους οποίους εκτιθέμεθα. Στον κατάλογο τον οποίο λοιπόν συντάσεις, Υπάρχει το θέμα της αντιμετώπισης με ισότιμο τρόπο όλων των κατηγοριών των πιστωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εσωτερικό μιας κατηγορίας πιστωτών υπάρχουν διαφορετικοί τύποι. Αναφέρομαι εδώ σε κάποιες ε, λιανικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι αν φανούμε εδώ πάρα πολύ προσεκτικοί θα πρέπει να το κάνουμε βλέποντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους θέλουμε να μετριάσουμε νομίζω ότι θα πρέπει βέβαια κάποιες κατηγορίες να, διαθέτουν, να διατρέχουν κινδύνους όπως αυτοί οι οποίοι είναι κάτοχοι ομολόγων μακράς διάρκειας. Δεν πρέπει εκεί να ισχύουν κρατικές εγγυήσεις. Τώρα, ε, για το πτωχευτικό δίκαιο Οι μεταφορές ε, ρευστότητας οι οποίες γίνονται στα πλαίσια μιας ε, τέτοιας διαδικασίας, ιδιαίτερα στην αρχή της διαδικασίας πτώχευσης. Ίσως θα πρέπει να δει κανείς τις προτιμησιακές περιόδους έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται σε μια περίπτωση όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, αλλά να υπάρχει δυνατότητα ε, αλλαγής της πορείας εφόσον αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό για τον πίνακα βαθμολόγησης αν θέλετε. Προφανώς για τους κινδύνους που παρουσιάζονται είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ κάθε ελεγκτική αρχή θα πρέπει ε, να το έχει υπόψη του. Δεν ξέρω αν ένα σύστημα θα έλεγα με κόκκινο και πράσινο χρώμα η πορτοκαλί χρώμα, δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα υπεραπλουστευτικό, ίσως να είναι λίγο υπεραπλουστευτικό. Σχετικά τώρα με τις απαιτήσει σε επίπεδο κεφαλαίων, εγώ κοίταξα το άρθρο 136 σχετικά με τη δυνατότητα των ρυθμιστικών αρχών. Προφανώς οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες εξουσίες, αλλά η οδηγία στο 136 δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Εμείς θα θέλαμε να μην ζητάμε να υπάρξει κρατική παρέμβαση όταν υπάρχει μια μικρή παραβίαση σε έναν περιορισμένο τομέα, σαν παράδειγμα. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν σχετικά με, την οδηγία για τις απαιτήσει σε κεφάλαιο και σε ρευστότητα των τραπεζών και πώς εφαρμόζεται όταν έχουμε να κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, να αντιδράσουμε με διαφορετικό τρόπο απέναντι στα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει από τη μία μια παγκόσμια τράπεζα μεγάλου μεγέθους και από την άλλη μια μεσαία ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Φερέιρα, ε, Σάιρα μάλλον, για την εργασία της που είναι πολύ καλή βάση ανάλυσης. Αλλά επίσης θα ήθελα να αναφέρω και εγώ μερικά θέματα που θα έπρεπε να τα ξαναδούμε. Η χώρα μου το Λουξεμβούργο επλήγει πάρα πολύ από την χρηματοπιστωτική κρίση του 8. Έχουν πτωχεύσει τράπεζες, έχουν σώσει την δεξιά, την τράπεζα δεξιά δηλαδή. Και χρειάστηκε να ληφθούν και άλλα επίγοντα μέτρα σε διαμεθοριακή μεν βάση, αλλά άλλα όχι. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη, περισσότερη εναρμόνιση και να υπάρξει ένα γενικότερο πανενοσιακό πλαίσιο λύσης των τραπεζικών κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι έδρες των τραπεζών και οι θηγατρικές των τραπεζικών ομίλων θα την χάνουν ίσης μεταχείρισης. Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα η κρίση του 2008 το έδειξε. Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αντιδρούν σαν αντλίες, φέρνουν δηλαδή ως το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια από τις θηγατρικές τους προς την έδρα τους. Αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο φαινόμενο. Αν όμως υπάρξει πτώχευση κάποιου μήλου, πράγμα που συνέβη, και δεν αποκλείεται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο δυστυχώς, τότε τα κεφάλαια των αρχικών τραπεζών και των θηγατρικών τους εξαφανίζονται. και μόνον οι πιστωτές της έδρας μπορούν να ελπίζουν ότι θα τους επιστραφεί ένα τμήμα των κεφαλαίων τους. Αυτό αποτελεί πραγματικά άνηση μεταχείριση και είναι άδικη μεταχείριση. Το είπε και η κυρία Χιούμπνερ. Και όταν συστήνει η κυρία Φερέρα ίση μεταχείριση των καταθετών μεταξύ χωρών μελών πρέπει νομίζω να απαιτήσουμε επίσης και να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σε περίπτωση πτώχευσης τραπεζών που να θεωρεί τον τραπεζικό όμιλο στο σύνολό του με τις θρηγατρικές του σαν έναν ενιαίο οργανισμό χωρίς να διαχωρίζει το κέντρο από τις θηγατρικές. Κατ' εμέ είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και με ικανοποίηση άκουσα ότι και άλλοι βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Άλλο θέμα τώρα. Χρειάζεται ή όχι πλήρης εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μήπως κανένα άλλο χωριστό καθεστώς που να υποκαθιστά τα εθνικά μέτρα για περίπτωση αντιμετώπισης κρίσεων. Δεν έχω σίγουρη απάντηση, αλλά το βέβαιο είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πτώχευσης. Τώρα για τις θεσμικές τράπεζες, που, θέμα που αναφέρθηκε από άλλους, εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Και η κυρία Χιούβνερ το είπε. Ο διαχωρισμός μεταξύ θεσμικών και μη θεσμικών τραπεζών ίσως να μην είναι ευκταίος. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι χρήσιμος. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε με βάση ποια κριτήρια θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Όλα αυτά είναι πολύπλοκα. Αν πάμε προς τα Κύπρο, στον τον διαχωρισμό δηλαδή, τότε θα καταλήξουμε σε μία νομοθεσία για τις θεσμικές τράπεζες και άλλη νομοθεσία για τις τράπεζες που θα έχουν διαμεθοριακές δραστηριότητες. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο. Εξάλλου, σχεδόν κάθε τράπεζα έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Άρα να ζητήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να εφαρμόζεται σε όλες τις διαμεθοριακές τράπεζες. Νομίζω ότι θα είναι λογικότερο κάτι τέτοιο και απλούστερο. Και τέλος, η μονάδα αυτή που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα πτώχευσης, η ρευτότητας, στην έκθεση της κυρίας Φεραίρα ζητάμε να δημιουργηθεί μια ειδική μονάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Και εδώ αναρωτιέμαι αν είναι σωστό κάτι τέτοιο. Η πτώχευση μιας τράπεζας είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και κακής εκτίμησης των εποπτών ή επιθεωρητών. Το είδαμε και κατά την ακρόαση του κυρίου Κωνσταντσα. Πρέπει λοιπόν σε όσους έχουν πτωχεύσει να δώσουμε τη δυνατότητα να ελέγχουν εκείνη τη ρευστότητα των τραπεζικών ομήλων. Το λογικό θα ήταν να προβλέψουμε έναν ανεξάρτητο οργανισμό ή κάποιο, κάποια διοικητική θέση να προβλεφθεί που ακόμη δεν υπάρχει. Έτσι θα αποφευχθούν ίσως και αντικρουόμενα, προβλήματα αντικρουωμένων συμφερόνιντων. Ευχαριστούμε πολύ υπερβάνς. Το κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Ελίζα Φερέρα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι πολύ χρήσιμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στιγμή που συζητάμε και με άλλες πλευρές τις οποίες σημείωσε στην εισαγωγή της, το πακέτο επίβλεψης δηλαδή. Είναι χρήσιμο να ασχοληθούμε και με το λεγόμενο αυτό τρίτο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο το οποίο έχει, θα έλεγα, υπογραμμιστεί ήδη από τον Τελαροζιέρ, όταν ήταν υπεύθυνο ε, μετά από απόφαση του Προέδρου Μπαρόσο. Αν θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί πραγματικά και καλά, θα έπρεπε να ξέρουμε τι συμβαίνει σε περίπτωση κρίσης. Όχι ότι θα πρέπει το σύνολο αυτής της πρόβλεψης διατάξεων να αφορά μία περίπτωση κρίσης, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα γίνει σε μια τέτοια περίπτωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε πολλά πράγματα για να πορευθούμε και καλό είναι να ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση. Τα θέματα είναι τόσο αλληλοσυνδεδεμένα που, αλληλοσυνδεδεμένα που δεν μπορώ παρά να εκφράσω μια ανησυχία όταν εκφράζει αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αναφερόμαστε σε μία ιδέα, κάθετα θα έλεγα, μία την ημέρα και προσπαθούμε να την κάνουμε να λειτουργήσει. Αλλά σε κάποια φάση θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση, θα πρέπει να υπάρξει μία διαιτησία. Οι τράπεζες δεν αγαπούν την πρόταση που λέει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα ίδια κεφαλαία τους. Αν δεν το δέχονται αυτό, τότε θα πρέπει να δεχθούν να τροφοδοτούν ένα ταμείο σταθερότητας η επίλυσης και αντιμετώπισης εν πάση περιπτώσει των δυσκολιών ε, στην περίπτωση που βρεθούν σε με τέτοιες δυσκολίες. Αυτό δεν το συζητάμε. Και αυτό είναι μια βασική ανησυχία που έχω. Μου λένε ότι η ομάδα των 20 θα ασχοληθεί με αυτό. Ναι εντάξει, αλλά Ξέρουμε πολύ καλά ότι με τα συμπεράσματα της ομάδας των 20 είναι μεν παίρνουν αποφάσεις αλλά μετά πάει ο καθένα σπίτι του και ασχολείται ελάχιστα με αυτά που έχει αποφασίσει. Νομίζω λοιπόν ότι τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινάει τη συζήτηση γύρω από το πρόβλημα επίλυσης των κρίσεων θα πρέπει να εντοπίσουμε ότι τα δύο αυτά πράγματα συνδέονται. Δηλαδή ή οι τράπεζες θα δεχθούν να ενισχύσουν σε βάθος την αυτορύθμισή τους αν θέλετε, οπότε σε αυτή την περίπτωση να αποφεύγουν τις κρίσεις ή να, όταν υπάρχει μια κρίση να είναι λιγότερο εκτεθειμένες και να υπάρχει ένα ταμείο διάσωσης, ε, αλλά αν δεν θέλουν να έχουν ίδιους πόρους τέτοιους ίδια κεφάλαια τα οποία θα τους δημιουργήσουν υποτίθεται προβλήματα ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αμερικανικά πιστοτικά συστήματα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δεχθούν να μπουν στη συζήτηση της δημιουργίας ενός ταμείου διάσωσης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο να επανέλθω σε μία σκέψη την οποία έκαναν πολλοί συνάδελφοι και την οποία συμμερίζομαι. Το πρόβλημα δηλαδή του τι είναι μία θεσμική τράπεζα ή συστημική τράπεζα ή μεγάλη και σημαντική τράπεζα. Είναι το ερώτημα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια ιδέα η οποία προήλθε από έναν κατάλογο τον οποίο είχε δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το ξέσπασμα της κρίσης όπου υπήρχαν 40 ε, συγγνώμη, τράπεζες πιο σημαντικές από τις άλλες. Αλλά η κρίση έδειξε ότι δεν προέρχεται συστηματικά από αυτές τις δομές η κρίση. Και η Ισλανδική περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά. Και το Ιρλανδικό κράτος, το Ισλανδικό κράτος μάλλον. Υπάρχουν ε, δηλαδή γεγονότα σε μία χώρα που δημιουργούν κινήσεις κεφαλαίου που δεν συνδέονται καθόλου με τον διαμεθοριακό χαρακτήρα των δομών που συζητάμε, αλλά που οι κινήσεις αυτές υποχρεωτικά οδηγούν σε ε, προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος διασυνοριακές. Mm. Έχει σημασία να δει κανεί αν η τράπεζα που ξεκινάει τη διαδικασία αυτή δραστηριοποιείται σε 15 χώρε βέβαια, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Και εκεί η διαφοροποίηση ανάμεσα σε θεσμική, συστημική ή ό,τι άλλο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σχετικά τώρα με το dashboard, το πίνακα ελέγχου ή πίνακα αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ριζοσπαστικοί όταν συζητάμε για τα θέματα αυτά και ελπίζω η συγγήτριά μας να μπορέσει να πιέσει περισσότερο και προς την κατεύθυνση της, εργα... επεξεργασίας και της συγκροσιμότητας. Είναι το λεγόμενο τεστ κοπόσεως. Ο καλύτερος τρόπος, εφόσον πιστεύουμε, εν πάση στα τεστ κοπόσεως, στα stress test ε, είναι λέμε προτιμότερο ή πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους πίνακες αποτελεσμάτων αλλά να ελέγχουμε πραγματικά την ικανότητα της τράπεζας να αντιμετωπίσει πιέσεις. Τώρα στην εναρμόνιση σε περίπτωση πτώχευσης. Εδώ υπάρχει μια τεράστια φυσικά συνένεση αν και η προσπάθεια <clears throat> δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη. Δύο παρατηρήσεις στα πέση αυτού του πάζλ που έχουμε μπροστά μας και όπου οι διαιτησίες αν θέλετε, οι προσπάθειες συμβιβασμού δεν δείχνουν να αποδίδουν. Εγώ σαν συνεισηγήτρια έχω κάποιες ανησυχίες. Αν εξετάζουμε κάθε φορά μια νομοθετική ρύθμιση με ένα συγκεκριμένο στόχο, ξεχνάμε τον βασικό μακροπρόθεσμο στόχο που είναι η ασφάλεια των επενδύσεων γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα πλαίσια των προτάσεων που ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε αυτή τη φάση, υπάρχει από τη μία το Ταμείο Σταθερότητας των Μεγάλων Τραπεζών, το οποίο τίθεται κινδύνο, από την άλλη όμως υπάρχει και η, ιδέα του Ταμείου εγγύ, ή μάλλον των εγγυήσεων των συστημάτων κατάθεσης, καταθέσεων θα πρέπει να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή για να δούμε σε ποιο βαθμό οι τράπεζες να μας πούν ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο. Η εναρμόνιση πάντως και ο ευρωπαϊκός καθορισμός ενός συστήματος εγγυήσεων των καταθέσεων έχει ενδιαφέρον. Σας θυμίζω Πρόεδρε ότι όταν, πως όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρυσι αν θυμάμαι καλά, αυξήσαμε τα ανώτατα όρια εγγυήσεων για τις καταθέσεις, είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προβλέψουμε ένα σύστημα, θα έλεγα, εναρμονισμού αυτών των εγγυήσεων των καταθέσεων. Έχει μεγάλη σημασία να γίνει κάτι τέτοιο. Σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτού του Ταμείου Σταθεροποίησης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ένα τέτοιο ταμείο να μην ευνοήσει τις ε, τράπεζες καταθέσεων αποκλειστικά και να θίξει τις δραστηριότητε κινδύνου, αυτές οι οποίες από την άλλη προκαλούν τους λεγόμενους διαμεθοριακούς συστημικούς κινδύνους. Οπότε η τροπή απόδοσης ε, ε, και οι τρόποι γενικά προσπάθειας κέρδους και κερδοφορίας θα πρέπει να επανεξεταστούν. Εντάξει, ο Πέτρος. Ευχαριστώ την Ελίσσα για την εξαιρετική της έκθεση και τις προσπάθειες που έκανε. Είναι προφανές ότι μια τέτοια έκθεση τη χρειαζόμασταν και βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια Βλέπετε βέβαια ήδη από τις αντιδράσεις ότι πολλοί θα ζητήσουν αντιφατικά πράγματα, αλλά αυτά που είπε η φίλη μου η Περβάνς, νομίζω ισχύουν και για τις πτωχεύσεις. Υπάρχουν όντως διαφορετικά συστήματα λειτουργίας επιχειρήσεων και τραπεζικών λειτουργιών ανάλογα με τις χώρες και επειδή πρόκειται για τεράστια κεφάλαια πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Υπάρχει ο φόβος να βιαστούμε και να μην λάβουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές που πρέπει να αναλύσουμε για να πετύχουμε τη σταθερότητα. Αλλά βέβαια τώρα σήμερα μιλάμε ιδιαίτερα για τις τράπεζες. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα που μας δίνεται είναι πολύ σωστό νομίζω να γίνει πρόταση της Κομισιόν μέχρι τα τέλη του 2011 και να την επεξεργαστεί από εκεί και πέρα το Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει από σήμερα να νομίζουμε ότι ό,τι πούμε σήμερα θα εφαρμοστούν από του χρόνου. Αλλά πάντως οι γενικές ιδέες είναι εξαιρετικές. Πρέπει να ρωτήσω όμως το εξής. Ωραία. Ξέρουμε ότι οι τραπεζικές λειτουργίες ήταν ο λόγος, ο μεγαλύτερος λόγος της δημιουργίας των πρόσφατων προβλημάτων αλλά είναι, ισχύει το ίδιο και για τα αποτελέσματα της κρίσης. Νομίζω ότι ο λόγος είναι διαφορετικός από το αποτέλεσμα. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε λοιπόν στην προσέγγιση μας ποιες τραπεζικές λειτουργίες ήταν λόγος και ποιες ήταν αποτέλεσμα της κρίσης. και πρέπει επίσης το Κοινοβούλιο να συζητήσει τι θα κάνουμε με την έκθεση Φερέρα ως προς την ΕΣΜΑ, το ΕΜΠΑ και την τρίτη αρχή που θα δημιουργηθούν αρκετά γρήγορα. Γιατί πρέπει κάποτε να το δούμε και αυτό. Εγώ θα προτιμούσα να εφαρμοστεί το δικό σας χρονοδιάγραμμα να γίνει δηλαδή μια πραγματική συζήτηση και όχι μια βιαστική και πρόχειρη. Αν όμως δεχτούμε κάτι τέτοιο το τελευταίο, τότε τουλάχιστον να βασιστούμε στο ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα αποκλείσει τις τροπολογίες που θα μας υποχρεώνουν ως Κοινοβούλιο να δεσμευτούμε με τις τρεις αυτές αρχές και να δεχόμαστε ό,τι πουν εκείνες. Δεν πρέπει να δείξουμε ανευθυνότητα, αλλά να παίξουμε ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Για να μην φανεί ότι εγκρίνουμε την αλαζονία ορισμένων μεγάλων τραπεζών οι οποίες έχουν κεφάλαια τα οποία παίρνουν απλώς από άλλες τράπεζες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να το προσέξουμε. Τι είχε προτείνει ακριβώς η Ελίσσα. Ναι, ίση μεταχείριση θεσμικών και μη θεσμικών τραπεζών, αλλά και ο Αμερικανός ειδικό που είχε έρθει να μας μιλήσει είχε πει ότι τέτοιου είδους διαχωρισμούς μπορούμε να τους κάνουμε με βάση το παρελθόν, αλλά για το μέλλον δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Εδώ μιλάμε για διαμεθοριακές τράπεζες. Υπήρξε η περίπτωση της Ισλανδίας και οι τράπεζες των γερμανικών κρατηδίων και τίποτε από αυτά, από όσα μέτρα ελήφθησαν για αυτά, δεν θα μπορούσε να ισχύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει λοιπόν πράγματι να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να περιλαμβάνει η νομοθεσία που θα εγκρίνουμε πριν βιαστούμε να δεσμευτούμε με, οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε άλλους. Επίσης υπάρχουν τράπεζες σήμερα που δεν, ε, δεν έχουν αρκετά κεφάλαια στις χώρες όπου λειτουργούν και βασίζονται στα κεφάλαια του ομίλου τους γενικότερα, του κέντρου δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε και αυτό από τώρα, να μην το αγνοήσουμε. Και αν θέλουμε όντως εξισορρόπηση των ευθυνών της τραπεζικής λεγόμενης βιομηχανίας, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς προς τα που θέλουμε να κινηθούμε και με τι μόνιμα ή προσωρινά μέτρα. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Φερέρα. Η πρότασή της είναι μια καλή πρόταση. Περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία. Πρώτον νομοθετικά και ρυθμίσεις, ελεγκτικές διαδικασίες και αντιμετώπιση της κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια μιας κρίσης δεν μπορούμε να εμένουμε στην αυτορύθμιση. Απαιτούνται άλλοι μηχανισμοί. Και εδώ θα συμφωνήσω με τις προτάσεις τις οποίες κάνει η πρόταση αυτή. Θα πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι στην κρίση να προστατεύσουμε φυσικά τα συμφέροντα των καταθετών, των επενδυτών και των φορολογουμένων. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ότι κάποιοι ολίγοι θα επωφελούνται από το σύστημα αυτό και όλοι οι άλλοι θα πρέπει να τους καλύπτουν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε την ευθύνη που έχει κάθε ομάδα και να προσπαθήσουμε να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι ομάδες αυτές. Απαιτείται λοιπόν ένα πλαίσιο, απαιτούνται εναλλακτικέ λύσεις, πότε θα τεθούν σε εφαρμογή εναλλακτικέ αυτές λύσεις και να δούμε ακριβώς τι είναι αυτά τα τεστ κοπόσεως, τα stress test εν πάση Τώρα για τις λεγόμενες θεσμικές, συστημικές ή εν σημαντικές γενικότερα τράπεζες Πράγματι υπάρχουν τέτοιες τράπεζες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Αν αυτό το οποίο θέλουμε είναι απλά να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε αυτές τις τράπεζες, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε επί τη βάση μιας πολυμερούς μεθόδου, όπως ακριβώς το κάνει η ομάδα των 20, το G20. Μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στα πλαίσια αυτής της περίπτωσης, αλλά αυτό δεν αποκλεί την παγκόσμια διάσταση. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί, ας αποφύγουμε κάποιες μονομερείς διαδικασίες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν πρόορες. Θα πρέπει να αντιδράσουμε σε επίπεδο πολυμερές. Και αφού το κάνουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να προχωρήσουμε δηλαδή και στα δύο επίπεδα παράλληλα. Μιλάμε επίσης και για ένα ταμείο σταθερότητας. Δεν είναι το ίδιο με ένα ταμείο ασφαλείας των καταθέσεων βέβαια. Πάρα πολύ συχνά τα ταμεία δίνουν εγγυήσει για τις καταθέσεις και επιτρέπουν έτσι την αναδιάρθρωση του συστήματος το να αναδιαφρώσει κανείς μια τράπεζα είναι πιο απλό από το να επιστρέψει τα χρήματα στους καταθέτες στην τράπεζα αυτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο κοστίζει συστηματικά περισσότερα και μιας και υπάρχουν καταθετικές τράπεζες και τράπεζες επενδυτικές, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι οι επενδυτές είναι αυτοί οι οποίοι δεν προστατεύονται επαρκώς. Γι' αυτό ακριβώς και χρειάστηκε να προσφύγουμε σε διαφορετικά συστήματα προστασίας όπως το TBS. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προστασίας του επενδυτή έτσι ώστε να αποφύγουμε να υπάρχει πάντα κρατική εγγύηση σε περίπτωση κρίσης. πέραν τούτου θα πρέπει στην Ευρώπη να έχουμε πολλά επίπεδα θα έλεγα δυνατότητας παρέμβασης. και δεν θα πρέπει να συγχαίρουμε τους ρόλους. Μπορούμε να ζητάμε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σαν παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ίδια κριτήρια για την αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η συνάδελφος κυρία Ήπνερ που αναφέρθηκε στην έκθεση του ΟΣΑ. Και εγώ την είχα μελετήσει στην έκθεση αυτή. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ιδίω όσον αφορά τι αιτίε ε, τη κρίση και τι σχετικέ προτάσει. Η ΩΣΑ, όπω είπαμε, προτείνει να προχωρήσουμε τους δύο τομείς ε, των ε, θεσμικών και των εμπορικών τραπεζών. Αναφέρατε διάφορες τράπεζες που ήταν επιτυχής ε, με την μεθοδολογία που ακολούθησαν και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποιες ήταν, ποιοι ήταν ακριβώς οι λόγοι που οδήγησαν στην κρίση θα ήθελα να ζητήσω να συμπεριλάβουμε και αυτή την πτυχή. Γιατί στο κάτω-κάτω ΣΑ δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι ένα σώμα πάρα πολύ ε, έγκαιρο και που πρέπει να λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και το θέμα του μεγέθου των τραπεζών άμεσα έστω λαμβάνει υπόψη ότι εάν ε, οι τομεί διανεμηθούν κατά τέτοιο τρόπο σε αυτοί οι δύο τομεί να μην συνδέονται μεταξύ τους, τουλάχιστον όσον αφορά την ευθύνη που έχουν, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι η πρόταση αυτή έχει οπωσδήποτε σημασία έτσι Εγώ θα θέλω να πω ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την πτυχή και να τη λάβουν υπόψη μας στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίλβη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μου λοιπόν, που θέλω καθυστέρηση, ήμουν κάπου αλλού, αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση εξ μου και να μιλήσω και χρειαζόμαστε στο Όλη Σμιτ που με παρακάλεσε να πω κάποια λόγια. Αυτό που λέω τώρα εγώ προσωπικά είναι όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο. Γιατί έχουμε μάλλον τάση να θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να διαφρυνήσουμε με ακρίβεια το συστημικό αυτό κίνδυνο γιατί μπορούν να οδηγούσε σε ένα κενό της ε, νομοθεσίας πολύ επικίνδυνο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρω του συνάδελφο Σμιτ που δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα και ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διαφοροποίησης, γιατί νομίζω ότι όλες οι τράπεζες θα πρέπει να πάρουν στο ίδιο καθεστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φεραίρα για την εκθεσή της. Από εκεί ίσως θα έπρεπε να ε, ξεκινήσω, να τη πω ότι συμφωνώ και με την προσέγγιση τη που ζητά την Κομισιόν να, επιβά, ε, να υποβάλει μέχρι το 2011 ε, μια γραπτή πρόταση για τη διαχείριση της κρίσης, γραπτή πρόταση, και συμφωνώ να εξτάσουμε από κοινού τους κανόνες ε, της ε, χρεοκοπίας και της έλλειψης ρευστότητας. Είναι σημαντικό να μην επιβαρύνουμε τους ε, Φελογούμους και από ό,τι φαίνεται η Σουηδία έχει κάποιο σύστημα και από αυτού θα ήθελα να πω στην κυρία Φερέρα ότι συμφωνώ με τι κυρίε τη ε, παρατηρήσει. Δεν θέλω να επαναλάβω τα πάντα. Είναι πράγματι αλήθεια ότι είχαμε στην Επιτροπή κρίση μια ακρόαση για την Σουηδία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί οι Σουηδοί μπόρεσαν να περάσουν ικανοποιητικά από μια πάρα πολύ άσχημη κρίση στη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εδώ έχουν μιλήσει όλοι εκτός από μένα. Όπως και άλλοι θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την έκθεση της Ελίσσα. Ξέρω, όταν αρχίζει κανένας να εξετάζει το θέμα αυτό, καταλήγει σε περισσότερες ερωτήσεις από ότι έχει απαντήσεις. Και οι διαφυλέψεις με την Κομισιόν είναι σημαντικές. Ε, ήταν καλό που ήταν εδώ η η να σημειώσει και ιδίω στη σχολιά μου για την έλεξη ρευστότητα που δεν θέλω να επαναλάβω. Το δίλημα στο οποίο βρισκόμαστε είναι ότι χρειαζόμαστε να προσβλέπουμε στο μέλλον φιλόδοξα. Από την άλλη μεριά όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζητάμε μια γλίγορη διόρθωση τη κατάσταση. Και όπω είπε η Κομισιόν μέχρι τα τέλη του επόμενου έτου. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ γλίγορο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποια ισορροπία. Αν δούμε το θέμα της ε, μεταφοράς ε, και της δίκαιης μοναχής μεταξύ των ομάδων, είναι κάτι που ανέφεραν ε, ορισμένοι από συναδέλφους. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και πολλές φορές σκέφτομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο το θέτουμε ίσως δεν είναι απόλυτα σωστό. Όταν εγώ εργαζόμουν για, στο θέμα στρατηγίας 2 για την χρηματοδοτία, είχα <clears throat> την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρχει μια κατανομή των πόρων χρονικά εν ώψη μιας επικείμενης έλλειψης ρευστού. είναι σαν μια διαθήκη, ποιος θα πάρει τι δηλαδή όταν πεθάνετε και ένα θέμα σαν να πρόκειται για μια φορολογία στην περίπτωση αυτή. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι σωστό ότι θα πρέπει καταρχήν να εξεταστεί με ένα ειδικό καθεστώ για τις τράπεζες, γιατί αλλιώ θα έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα που και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και αν εξετάσουμε με τα πράγματα μακροπρόθεσμα, είναι γελίο να περιμένουμε να έχουμε ενιαία αγορά, εσωτερική αγορά, και να μην έχουμε επαρκούς ε, μηχανισμούς για την ενταμισόπιση χρεοκόπησες. χρεοκόπησης. Και αν μου επιτρέψετε τώρα να στραφώ προς το ταμείο στο οποίο αναφέρεστε, μάλλον θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ε, επιβολή κύρωση στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο σφαλμένα. ο οποίο θέλει να το χρησιμοποιήσει δηλαδή, θα πρέπει κάτι να υποστεί. Ε, τουλάχιστον εκείνοι που έχουν αναλάβει τους κινδύνους της τράπεζας πρέπει κάτι να αισθανθούν ότι συμβαίνει. Και η παρατήρησή σας για το ίδιο το ταμείο. Um, ε, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε νέο τύπου κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο σταθερότητας, η επίλυση κρίσης, όπως θέλετε πείτε το, θα μας βοηθήσει νομίζω από το να έχουμε πιο ξωτικές μορφές, αν μπορώ να τις πω έτσι, κεφαλαίου που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα εις βάθος και να μελετήσουμε κατά πόσον έχουμε εξετάσει και τι κάνει η Βασιλεία για το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να δημιουργούμε κάποια ξωτικά πράγματα και από την άλλη μεριά να λέμε όλα θα πρέπει να είναι πιο απλά. Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ταμείο τι μεγέθους θα είναι. Γιατί άμα δούμε το spread που υπάρχει στις ε, τράπεζες του Ρωμανού Βασιλείου βλέπουμε ότι η αξία των εγγύσεων είναι ίση με το όφελος που έχουν οι τράπεζες των 50 δισεκατομμυρίων νομίζω θέλουμε εκεί να κινηθούμε. Κάτι θα πρέπει δηλαδή, να γίνει πριν. Νομίζω ότι όσον αφορά αυτές τις διαθήκες, θα μπορούμε να τις πούμε έτσι, και τα διάφορα επιχειρήματα για το προς τα που θέλουμε να κινηθούμε ακριβώς, θα πρέπει νομίζω να παίρνουμε και μια δυνατότητα διαφυγής για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα θα εξακολουθεί να μπορεί να λειτουργήσει. Βέβαια υπάρχουν και διάφορες λύσεις που μπορούν να αποτύχουν. Εμείς δεν θα πούμε ότι αν κάτι είναι υπερβολικά μεγάλο για να το αφήσουμε να αποτύχει, θα το διαθώσουμε θα διασώσουμε ολόκληρο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Πάντως ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά και μας προσανατολίσατε πολύ ωραία όσον αφορά κάποια από τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε εδώ, πριν απαντήσετε, να πούμε ότι μια εδώ πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία. Υπάρχει μια πολύ αυστηρή δομή. Αυτοί που ήταν στην παρασμένη θητεία εδώ θα ξέρουν πώς, τι κάναμε την έκθεση Ράσμουσεν. Είχαμε ένα πρώτο τμήμα δηλαδή που έχει κάποιες ιδέες που προσανατολίζουν προς τα εμπρός. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να έχουν κάποιες πιο συγκεκριμένε συστάσεις όπου ζητάμε να υπάρχει νομοθεσία. Θα υπάρχει δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάτι. Τώρα έχουμε ένα νέο κανόνα διαδικασίας, ε, των κανόνα υπαριθμών 42, το άρθρο υπαριθμών 42 και η γραμματεία θα πρέπει να δει τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την μορφή παρουσίασης της οδηγίας. Αλλά νομίζω θα είναι κάτι παρόμοιο με εκείνο που είχαμε πετύχει με την έκθεση Rasmus. Αλλά θα σας το ανακοινώσουμε έγκαιρα πριν από την προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Καλό ήταν να το πω εδώ τώρα, νομίζω και να μην στο πω στο τέλος. Ελίσσα, δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε? Και επίση θα θέλαμε να προσπαθήσουμε να έχουμε για του συντονιστέ και λίγο χρόνο διερμηνίας αν είναι δυνατόν. Αν όχι, τι να γίνει. Well, Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, για τις ερωτήσεις, τις προτάσεις, την κριτική, την στήριξη. Έχω σημειώσει πάρα πολλά πράγματα που είπατε. Θα ήθελα να έχω και προσωπικές επαφές με όσους από εσά θα ήθελαν με συγκεκριμένο τρόπο να κάνουν προτάσεις βελτίωσης της προσπάθειάς μου. Πάντα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τόσο περίπλοκη δεν μπορούμε να επιλέξουμε αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε, αλλά προσπαθούμε να φανούμε συμβιβαστικοί και ρεαλιστές. Αυτή είναι η ουσία της προσπάθειας την οποία κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάθε μία από τις ε, ερωτήσεις, θα ήταν παράλογο. Σημείωσα όμως όσα είπατε για τις μεταφορές ρευστότητας Αυτό συνδέεται και με μια πολιτική επιλογή την οποία πρέπει να κάνουμε και να προωθήσουμε. Σε αυτή τη φάση ή θα ενισχύσουμε ό,τι έχει σχέση με την ισχύ της εσωτερικής αγοράς ή θα υπαναχωρήσουμε σε μια προστατευτική εθνική αντίληψη. Νομίζω ότι η πρότασή μου και η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά, ενίσχυση μάλλον της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε να μπορούμε και σε διεθνές επίπεδο να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Πέραν τούτου όμως, λαμβάνω υπόψη ότι υπάρχουν εθνικά συμφέροντα και εθνικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό προτείνω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη φάση εναρμόνισης μέσω της ενίσχυσης του συνόλου της ομάδας των ελεγκτών υπό την διεύθυνση θα έλεγα υπό τον ηγετικό ρόλο της EBA. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη λύση την οποία προτείνω μέσω της ε, <clears throat> ενημέρωσης και επικαιροποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης, εμπλέκοντας και τους Υπουργούς Οικονομικών, οι οποίοι προφανώς έχουν πολλά να πούν σε επίπεδο έκφρασης των εθνικών συμφερόντων. Το θέμα είναι να μην το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν κάτι το στάσιμο, αλλά σαν ένα τρόπο προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης κάθε οργάνου, του τρόπου με την μεθοδολογία που κάθε ε, ελεγκτική αρχή χρησιμοποιεί, για να αποφύγουμε τις καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε στις παρελθούσες κρίσεις, όπου κάποιες από αυτές τις αρχές συναντιόντουσαν σοβαρά για πρώτη φορά. Σε μια πολύ κρίσιμη φάση, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια σαφέστατη, εκεί υπήρξε μάλλον μια σαφέστατη έλλειψη συγκεκριμένης κατανόησης του ρόλου και του εύρους του συγκεκριμένου οργάνου, της ελεγκτικής αρχής δηλαδή. Τώρα για τις λεγόμενες συστημικές ή θεσμικές τράπεζες. Θα ήθελα να ενισχύσω την ιδέα να μην αντιμετωπίσουμε τις τράπεζες αυτές σαν μια εντελώς ανεξάρτητη ομάδα τραπεζών Θέλουμε εμείς να έχουμε ένα κοινό βιβλίο κανόνων, κοινή κατανόηση, μια ευρωπαϊκή συνολική αντιμετώπιση. Αν αρχίσουμε στη συγκεκριμένη φάση όμως να δίνουμε βασικά στην EBA τον ηγετικό ρόλο για τη διαχείριση των κρίσεων για όλες τις τράπεζες, τις διεθνείς, αυτό θα είναι παράλογο. Το θέμα είναι να δούμε αν όλες οι τράπεζες, ακόμα και αυτές οι τράπεζες οι διαμεθοριακές, θα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το Ταμείο Σταθεροποίησης. Αν τους ζητήσουμε να συνεισφέρουν σε αυτό το Ταμείο, τότε η διάσωση, η μη διάσωση θα πρέπει να προέλθει από τις συγκεκριμένες αυτές τράπεζες. Οπότε επανερχόμαστε στον ρόλο τον οποίο θα πρέπει να παίξει το EBA. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε φτάσει εκεί και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα είναι εφικτό να φτάσουμε σύντομα. Ένα τρίτο θέμα είναι ποιος είναι ο στόχος αυτής της παρέμβασης. Η Βίκη είπε ότι πράγματι μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσουμε μια τέτοια συστημική σε εισαγωγικά τράπεζα, αλλά αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα. Και θέτει εδώ και το πρόβλημα του μεγέθους του ταμείου αυτού. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο βασικός στόχος της έκθεσης, αλλά στην αιτιολογική έκθεση εγώ υπογραμμίζω ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι η δημόσια διάσταση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αποκατάσταση ή ευθανασία. Είναι δύο ξεχωριστές επιλογές. Αν επιλέξει κανείς την ευθανασία ή την αποκατάσταση, έχει, θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη αντίληψη για τη συγκεκριμένη περίπτωση το ποιος θα το πληρώσει. Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτές ακριβώς τις διασυνοριακές ε, επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκρινίζουμε το ποιος θα καλύψει το κόστος μιας τράπεζας επτόχευσης. Ποιος θα καλύψει την βοήθεια διάσωσης μιας τράπεζας που κινδυνεύει. Και το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ε, χαρακτηρίζεται από κοινού στόχους όσων συμμετέχουν. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης αυτό που είπε ο Σβέν στο σημείο 8, ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας το toolbox που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσφέρεται προς συζήτηση βέβαια. Από την άλλη δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε συστηματικά διαφορετικά τους καταθέτες και τους επενδυτές ανάλογα με τη χώρα και την εθνικότητά τους. Αυτό το είναι κάτι το οποίο επιμένω ήδη στο πρώτο μου σημείο. Πέραν όλων αυτών υπάρχουν και άλλα θέματα όπως το DGS, τα έκτακτα προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων, όταν μια μεγάλη τράπεζα μεγαλώνει και συνδέεται με πολλά χρηματοπιστωτικά συστήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη πρόταση, τι κάνουμε. Αυτό είναι μια δυσκολία. Το θέμα είναι πόσο μακριά μπορεί κανείς να φτάσει σε ένα πρώτο επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να φανούμε διαλλακτικοί και στα πλαίσια αυτής της συνδιαλλαγής εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο μπορούμε αλλά όχι πάρα πολύ μακριά γιατί τότε τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. <coughs> Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Θα λάβω υπόψη ό,τι είπατε και μπορώ να το εφαρμόσω στην πρότασή μου και φυσικά εφόσον θέλετε να γίνει πιο αναλυτική συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει σε μικρή κλίμακα είμαι στη διάθεσή σας. In this, in this present session. Uh, thank you very much to all of you and... Uh, είμαι στη διάθεσή σας. Περιμένω τις προτάσεις σας. Λοιπόν, έχουμε δικαίωμα. Ε, ευχαριστώ πολύ. For this is the deadline for the amendments is noon on. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι μεσημέρι 27 Απριλίου είναι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Θα τις εξετάσουμε την 1η Ιουνίου, τις επιλογές αυτές. Θα τις ψηφίσουμε στην Επιτροπή αυτή έκον στις 22 Ιουνίου και θα περάσουμε στην Ολομέλεια μετά τις ελληνές διακοπές για την πρώτη, στην πρώτη συνόδο του Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πρώτο χρόνο που προβλέπεται αυτή τη στιγμή και ελπίζω να μπορέσουμε να το τηρήσουμε. Εδώ ολοκληρώνουμε κατά βάση την συνεδρίασή μας. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα ήθελα να παραμείνουν οι ε, και άλλοι άμα θέλουν βέβαια να έχουμε δύο-τρεις κουβέντες για την ακρόαση της Τετάρτης το απόγευμα.